Dear colleagues, if you could please take... Παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. Good afternoon and welcome, colleagues, and, and welcome to our guests. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Σημείο πρώτο, έγκριση μερίσες διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, την εγκρίνουμε. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Καταρχήν, ε, διερμηνία. Δυστυχώς, δεν έχουμε διερμηνία ε, στα κροατικά, μαλτέζικα και γοεδελικά. Και θα πρέπει να εγκρίνουμε και τη στάση των συντονιστών ε, με βάση τον 205 ε, κανόνα. Καταρχήν, ο κ. Υγιασδόφσκι του ΕΛΚΑ ορίστηκε εισηγητή για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Νορβηγία για του συμπληρωματικού κανόνε για τα μέσα χρηματοδοτική υποστήριξη για τα εξωτερικά σύνορα και τι θεωρήσει. Στα πλαίσια του Ταμείου Εσωτερική Ασφάλεια για την περίοδο 2014-2020. Έχουμε δύο εισηγητέ για τι γνωμοδοτήσει. Ο κύριο Πίτερσον από την Άλτε, που ορίστηκε εισηγητή για τη γνωμοδότηση τη έκθεση των Σώμα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστών για τι Ελεκτρονικέ επικοινωνίε και ο κύριο Σόγκορ του ΕΛΚ ορίστηκε εισηγητής τη γνωμοδότηση για την έκθεση σε ό,τι αφορά το νέο εμπορικό πλαίσιο για τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία. Συμφωνείτε με τη στάση των συντονιστών. Μάλιστα. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών της 17ης Οκτωβρίου του 2016. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τα πρακτικά, θα τα εγκρίνουμε και αυτά. Περνάμε στο σημείο 4. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς πώς ε, θα διαρκέσουν τα διάφορα σημεία. Πρέπει να έρθουν πρώτα οι αρμόδιοι ομιλητές. Είναι αυτονόητο βέβαια αυτό που λέω. Περιμένουμε τον πρόεδρο Σούλτς. Θα καταφτάσει ένα πάση στιγμή. Ο καθηγητής Μπούντε είναι παρόν. Δεν ξέρω αν θα ήθελε να ανέβει στο βήμα. και ελπίζω να έρθει να πάσει στιγμή και ο πρόεδρος Σούλτς. Θα κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή εν αναμονή του Προέδρου για να μπορέσουμε να περάσουμε στο πρώτο σημείο, το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ για τη συνεργασία. Α, α συγγνώμη. Νόμιζα ότι εσείς ήταν ο καθηγητής Μπούντε. Ούτε και εκείνος έχει έρθει ακόμη. Ο καθηγητή Μπούντε είναι στο ίδιο αυτοκίνητο με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οπότε θα έρθουν μαζί μια δίλεπτη διακοπή και μόλις έρθουν οι καλεσμένοι μας θα ξεκινήσουμε. So, Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Οπότε, περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσης διάταξης, στη χάρτα ε, θεμελιωδών ψηφιακών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρθουν, έχουν έρθει στο μεταξύ καλεσμένοι μας. Η, παρουσίαση θα γίνει παρουσία του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κ. Μάρτιν Σούλτσε, από τον καθηγητή Χάιντ Πούντε, από την ομάδα των συντακτών αυτής της χάρτας θεμελιωδών ψηφιακών δικαιωμάτων. Έχετε λάβει ε, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τον χάρτη αυτό και ελπίζω να τον έχετε κοιτάξει. Υπάρχουν και μερικά αντίγραφα σε χαρτί στην αίθουσα. Όσοι δεν γνωρίζουν το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου, τη Χάρτα των Θεμελιωδών Ψηφιακών Δικαιωμάτων, καταρχήν να καλωσορίσω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είστε ευπρόσδεκτο στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, κύριε Πρόεδρε. Θα έχουμε εδώ τα εγγένεια αυτού του χάρτη που είναι το απάβγασμα μιας διεπιστημονικής ομάδας ε, καθηγητών ε, νομικών, πολιτικών, ε, blogger, δημοσιογράφων και έχει δημοσιευθεί σε πολλές έγκριτες εφημερίδες, Zeit, Welt, Welt Compact και ούτω καθεξής. Και ε, η Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή είναι εξοικειωμένη αυτό το θέμα και μάλιστα και ο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρακολουθεί από την αρχή το θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με ιδιαίτερη χαρά και εγώ και οι συντονιστέ τον καλωσορίζουμε και την πρώτη παρουσίαση, την επίσημη παρουσίαση αυτού του εγγράφου. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον Πρόεδρο Σούλ και στον καθηγητή Μπούντε από την ομάδα των συντακτών αυτού του χάρτη θεμελιωδών ψηφιακών δικαιωμάτων για να μα κάνουν μια σύντομη εισαγωγή και μετά συνάδελφοι θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλλετε τα σχόλιά σας ή να θέσετε τις ερωτήσεις και τις απορίες σας. Μάρτιν, έχει το λόγο και σε ευχαριστούμε θερμά που ήρθες. Κλοντ, Ευχαριστώ. Κλοντ, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε. Η παρουσία του Προέδρου σε μια επιτροπή είναι, είναι μια πρωτοφανής λίγο πολύ διαδικασία στην, ε, θη, θητεία μου τουλάχιστον ως Προέδρου του Κοινοβουλίου είναι η πρώτη φορά που παρίσταμε σε συνεδρία της Επιτροπής και αυτό οφείλεται στο θέμα. Γιατί θέλω με την παρουσία μου να τονίσω πόσο σημαντική είναι για μένα η εκπόνηση ενός χάρτη θεμελιωδών ψηφιακών δικαιωμάτων εδώ στην Επιτροπή Ατομικών Ελευθεριών και Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. συμμετοχή λοιπόν του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια τέτοια ε, ε, επιτροπή, συνεδρίαση επιτροπής ε, οφείλεται σε ιδιαίτερους λόγους όπως είπα και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω Κλώτη για το γεγονός ότι μου δίνεις το λόγο εδώ στην έναρξη αυτής της συζήτησης. Πριν από αρκετά χρόνια, όχι μόνο εδώ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ε, Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς μπορεί ε, η νομοθεσία γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων που αποτελεί τμήμα της ε, συνθήκης της Λισαβόνας πώς λοιπόν μπορεί ε, αυτά τα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην εποχή, ε, στην ψηφιακή εποχή να προστατευθούν σε μια περίοδο όπου ενδεχομένως ε, κινδυνεύουν ή απειλούνται. Πώς μπορούν αυτά τα δικαιώματα να εξασφαλιστούν ε, και σε έναν ψηφιακό κόσμο. Ασχοληθήκαμε πολύ με αυτό το θέμα και αποφασίσαμε, καταλήξαμε ε, αν θα μπορούσε, ε, ε, ότι θα, έπρεπε να συμπληρωθεί ή αν θα ήταν δυνατόν να συμπληρωθεί η ισχύουσα χάρτα με μια επιπλέον χάρτα για τα ψηφιακά θεμελιώδη δικαιώματα. Αν θα ήταν, αν θα ήταν δηλαδή η κατάλληλη επιλογή να συμπληρωθεί ή να συνταχθεί μια νέα χάρτα Βάση και λόγω και των ε, ραγδαίων εξελίξεων ε, που συνοδεύουν αυτήν την ψηφιακή επανάσταση. Αυτό το ερώτημα λοιπόν από, διάφορα, από διάφορες κοινωνικές ομάδες ε, απασχόλησε μια ομάδα ανθρώπων και στο πλαίσιο αυτής της ομάδας εκπρόσωποι διαφόρων κοινωνικών ομάδων, διαφόρων ιδεολογικών ρευμάτων, οργανώσεων που είχαν ε, τη διάθεση να συζητήσουν και να συμμετάσχουν σε μια τέτοια διαδικασία. Συζήτησαν λοιπόν για πολύ καιρό και κατέληξαν στο αποτέλεσμα που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα εδώ. Εγώ προσωπικά συμμετείχα σε αυτές τις συζητήσεις, σε αυτή τη διαδικασία και το έκανα αυτό γιατί είμαι μέλος της ε, Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ξεκινήσαμε το έτος 2000 τη διαδικασία για τη σύνταξη για ε, του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ήμουν εισηγητής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και από τότε μάλιστα είχαμε συνεργαστεί με τον συνάδελφο Κάρλος Κοέλο ως ε, μέλος λοιπόν εκείνου του, ε, εκείνου του χάρτη για τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, παραμένω στις επάλξεις όσον αφορά το μέτωπο αυτό και τα τελευταία χρόνια με απασχολεί πολύ το ερώτημα σε ποια κοινωνία θέλουμε να ζούμε, πώς η ψηφιακή επανάσταση επηρεάζει την καθημερινότητά μας, την καθημερινή μας ζωή. Τον συνάδελφο Άλμπρεχτ που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής σας ε, συμμετείχε επίσης σε αυτήν την ομάδα εργασίας και το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε ε, θα σας παρουσιαστεί σήμερα εδώ. Χαίρομαι πολύ που μας δίνετε αυτή την ευκαιρία, αγαπητοί συνάδελφοι, και μιας και στη Γερμανία έχει ήδη προηγηθεί μια πολύ έντονη συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα, θα ήθελα να κάνω μια διαπίστωση. Κατανοώ τους ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τον εσωτερικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά αυτό που κάνουμε σήμερα δεν είναι μια νομοθετική διαδικασία, αλλά η παρουσίαση μιας ιδέας σε μια επιτροπή νομοθετική, αν θέλετε. Πρόκειται δηλαδή με άλλα λόγια για ένα βήμα με την ελπίδα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και άλλα όργανα και τα εθνικά κοινοβούλια θα ασχοληθούν με αυτό το ερώτημα της εκπόνησης της σύνταξη μια χάρτα ψηφιακών θεμελιωδών δικαιωμάτων και με το ερώτημα το πώς μπορούμε να ε, εξασφαλίσουμε, να εγγυηθούμε τα ψηφιακά δικαιώματα, ενδεχομένως να τα εμβαθύνουμε και να τα επεκτείνουμε. Να υπάρξει λοιπόν μια όσο το δυνατόν ευρύτερη συζήτηση. Αν ε, θέλετε λοιπόν και επειδή ε, δεν ε, είναι δεδομένο ότι οποιοδήποτε ασχολείται με αυτά τα ερωτήματα γνωρίζει και τα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να πω ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια τυπική νομοθετική διαδικασία. Θέλουμε να κάνουμε μια πλατιά συζήτηση γύρω από τα ζητήματα ε, που μας απασχολούν ως πολίτες για το αποτέλεσμα αυτό, ε, αυτόν που, ε, στο οποίο καταλήξαμε εμείς ως αποτέλεσμα στις συζητήσεις μας στην ομάδα εργασίας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και θα ήθελα κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας, ο κύριος Μπούντε να είναι εκείνος που θα σας παρουσιάσει το περιεχόμενο αυτής της ε, δουλειάς. Ο κύριος Μπούντε. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί λοιπόν μιλούμε για ψηφιακά θεμελιώδη δικαιώματα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το, ε, ο 18ος αιώνας ήταν ο αιώνας των ε, αστικών ελευθεριών, ο 19ος αιώνας ήταν ε, ο, ε, ο ε, ο αιώνας για την ε, συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες και ε, ο 20ος αιώνας των, ο αιώνας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε λοιπόν να ασχοληθούμε με το θέμα της χρήσης και της εφαρμογής των ψηφιακών δικαιωμάτων. Των δικαιωμάτων δηλαδή των ανθρώπων στην ψηφιακή εποχή. Πρόκειται στην ουσία για μια νέα βαθμίδα. Ας μην ξεχνούμε ότι σήμερα ζούμε όλοι σε μια ψηφιακή σφαίρα με την οποία ερχόμαστε σε καθημερινή επαφή, η οποία μας δίνει νέες δυνατότητες διαδραστικής ε, δικτύωσης, της ε, συνεργασίας, αλλά και της προσφοράς νέων ε, δυνατοτήτων. Και το ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι αν αυτές οι, αυτές οι νέες περιστάσεις αποτελούν ή επιφέρουν νέες δυνατότητες, νέες ελευθερίες ή και απειλές για τις ελευθερίες μας. Είναι σίγουρο ότι έχουμε να κάνουμε με ένα νέο τύπο ε, προκλήσεων, ε, προσφορών, ε, κάτι που θέτει και το ερώτημα τι, είναι τα, τι, τι είδους εμπορεύματα είναι τα δεδομένα με τα οποία έρχομαστε σε επαφή. Πρόκειται για καθαρά ιδιωτικά εμπορεύματα, ιδιωτικής ιδιοκτησίας ή υπάρχουν και δημόσιου χαρακτήρα δεδομένα. Τίθεται και το ερώτημα ποια θα είναι η χρήση αυτής της ψηφιακής σφαίρας, κάτι που συνδέεται και με το ερώτημα ποια είναι, ποιες είναι οι ευκαιρίες για τις ελευθερίες που θα έχει αυτή η νέα περίοδος. Το συζητήσαμε, το είπε και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ότι η ομάδα η οποία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα δεν είναι ομάδα εμπειρογνωμόνων. Ήταν μια ομάδα με μεγάλη ε, ποικιλομορφία. Υπήρχαν άνθρωποι από το διαδίκτυο, ε, δημοσιογράφοι, νομικοί, επιστήμονες της επικοινωνίας, ακτιβιστές ε, για τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά και διανοούμενοι όπως εγώ που συνήλθαν και συζήτησαν τα ερωτήματα. Τα ερωτήματα μας απασχόλησαν ήταν ποια είναι αυτά τα δικαιώματα ε, που χρειαζόμαστε στην εποχή μας και για την εποχή μας. Ήταν ξεκάθαρο σε μας ότι το κάνουμε, ε, κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά ιδίως για μια γενιά για την οποία το ψηφιακό αποτελεί αυτονόητη υποδομή η οποία ε, δεν θεωρεί ότι πρόκειται για κάτι για το οποίο χρειάζεται κάποιος ενθουσιασμός, αλλά το παίρνει ως δεδομένο. Πώ λοιπόν, και αυτό είναι το κύριο ερώτημα που θα έπρεπε να μας αποσχολήσει και από πολιτική σκοπιά. Πώς με ποια λόγια, με ποια διατύπωση, με ποια υλικά στοιχεία και με ποια στάση της κοινή γνώμης μπορούμε ε, τους digital natives αλλά και εκείνους που θα μάθουν τις ψηφιακές δεξιότητες εκ των να ε, χειριστούν τις ε, ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Από 1η Δεκεμβρίου, από τότε δηλαδή το είπε και ο πρόεδρος που δημοσιεύτηκε σε γερμανικές εφημερίδες και στο διαδίκτυο το κείμενο αυτό, ξεκίνησε μια αρκετά ζωηρή συζήτηση στο διαδίκτυο που... Ε, που απαιτεί ε, και θέτει ορισμένα ζητήματα για τους συντάκτες αυτού του κειμένου. Ο τίτλος ε, μάλιστα είναι ε, αμφιλεγόμενος. Για ποιον λόγο χρειαζόμαστε ψηφιακά θεμελιώδη δικαιώματα. Έχουμε και αναλογικά θεμελιώδη δικαιώματα. Δεν είναι έτσι και αλλιώς αδιέρετα τα, δικαιώματα αυτά στην ψηφιακή εποχή από τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα που έτσι και αλλιώς ισχύουν. Μήπως είναι θέματα όπως η πυρηνική ενέργεια που, που θέτει νέα ζητήματα, αναδεικνύει νέα προβλήματα. Θέλω να, να αναφερθώ σε ένα ζήτημα. Η λογοδοσία και η ευθύνη που έχουν οι μηχανές που λαμβάνουν αποφάσεις, κάτι που ε, ε, επηρεάζει όχι μόνο το ίντερνετ αλλά και την ίδια τη δημοκρατία. Και μετά είναι και το ερώτημα, το οποίο συζητήσαμε έντονα. Η διασύνδεση των ε, δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της αυτοδιάθεσης η αρχιτεκτονική λοιπόν ε, που, ε, με την οποία διαρθρώσαμε αυτόν τον χάρτη των ψηφιακών θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι η κατάλληλη, είναι η, είναι η ενδεδειγμένη. Τα, τα θέματα ε, δεν συνδέονται αυτά τα ψηφιακά δικαιώματα με, με δικαιώματα εμπιστευτικότητας και απορρίτου. Τρίτο, πολύ σημαντικό στοιχείο. Τι σημαίνει αυτή η νέα κατάσταση με την οποία με την οποία έχουμε να κάνουμε. Όσον αφορά το ερώτημα μιας νέας μορφής ιδιοκτησίας στην οποία συμμετέχουν οι δημιουργοί, οι παραγωγοί και οι χρήστες. Και ένα θεμελιώδες ερώτημα μας απασχόλησε επίσης τι σημαίνει, τι σημαίνει όταν παρουσιάζουμε ε, μια ιδέα για αυτήν την, ε, ε, για αυτήν την ε, νέα εποχή. Όταν τελειώσει δηλαδή αυτή η φάση της αρχικής συσσόρευσης, για να μιλήσω λίγο μαρξιστικά, τίθεται το ερώτημα μήπως θα έπρεπε να ε, έχουμε και ένα Υπουργείο Αλήθειας και Επαλήθευσης το οποίο θα ελέγχει τους αλγορίθμους Μήπως τελικά είμαστε οι λογοκριτές, οι, εκείνοι οι οποίοι θα περιορίσουν τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζουμε ότι τα, ερωτήματα και οι απαντήσεις που θα δοθούν θα διαμορφώσουν φυσικά και το χαρακτήρα και τη μορφή του τελικού αποτελέσματος. Αλλά θέλουμε να γίνει αυτή η συζήτηση. Γιατί θέλουμε να θέσουμε ενώπιον της κοινωνίας όλες αυτές τις προβληματικές, όλα αυτά τα ερωτήματα και θέλουμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ώστε η κοινωνία στην οποία ζούμε να, αρχίζει, να αρχίσει να ηχνηλατεί τη δική της πολιτική βούληση του πώς δηλαδή θέλει η ίδια να παρέμβει με δικαιώματα σε αυτήν την νέα ψηφιακή εποχή αν θέλει να την συνδιαμορφώσει ή αν ε, αντιθέτως θέλει να ε, αγνοήσει αυτή τη διαδικασία και να ε, λειτουργήσει ως απλός παρατηρητής. Αυτό που θέλουμε, θέλαμε δηλαδή με αυτόν, και θέλουμε με αυτόν τον χάρτη να, να επιτύχουμε είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία στο τέλος της οποίας θα εκφραστεί μια πολιτική βούληση της κοινωνίας κάτι που ενδεχομένως να ξεπερνά και τις δικές μας δυνατότητες αυτά που μπορούμε στο σήμερα να προβλέψουμε. Αυτά ως προς τον χάρτη από μένα έτσι εν συντομία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούντα. Αυτή η Επιτροπή έχει εμπλακεί εκτενώς αυτό το θέμα. Είχαμε και την έκθεση για την μαζική παρακολούθηση και γι' αυτό προσπαθήσαμε να ετοιμάσουμε τη χάρτα. Αλλά εδώ αποκρισταλώσατε διάφορα βασικά σημεία και οι συνάδελφοι έχουν κάποια σχόλια στα οποία θα ήθελαν να προβούν και ίσω κάποιε ερωτήσει. Πέντε συνάδελφοι επιθυμούν να λάβουν το λόγο Ιωσδήποτε οσδήποτε α το ζητήσει. Αλλά αν είμαστε ακόμα πέντε συνάδελφοι, ένα-δύο λεπτά ο καθένα έχουν το λόγο. Κύριε Χολμάια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπούντε, Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσίασή σας αλλά και για τις προσπάθειες που έχετε καταλάβει για να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση. Εγώ προσωπικά ε, ε, τηρώ κριτική στάση απέναντι σε ένα τέτοιο χάρτη ψηφιακών θεμελιωδών δικαιωμάτων γιατί έχουμε την, ε, τον, τον χάρτη για τα θεμελιώδη δικαιώματα που κανονικά θα έπρεπε και θεωρώ ότι πρέπει να καλύπτουν αυτά που αναφέρετε εσείς και μάλιστα τη συντάξαμε αυτή τη χάρτα σε μια εποχή που υπήρχαν ζητήματα τα οποία δεν είχαν ανακύψει ακόμα και τα οποία κληθήκαμε να απαντήσουμε, να, να απαντήσουμε στην πορεία δηλαδή ελευθερία ε, ε, αξιοπρέπεια, όλα αυτά είναι ζητήματα που ε, καλύπτουν και το διαδίκτυο. Για μένα πάντως το βασικό ερώτημα, ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι το εξής. Έχουμε τα big data, τα μεγάλα δεδομένα. Τι θα τα κάνουμε. Γιατί το να ευχόμαστε ότι θα εξαφανιστούν δεν θα μας, φέρει, δεν θα μας οδηγήσει κάπου. Ίσα ίσα τα υπόλοιπα τμήματα του κόσμου μπορεί και να χαρούν. Γιατί ακριβώς θα κατακτήσουν νέα μερίδια στην αγορά. Οπότε πρέπει εμείς να δούμε πώς θα επιβάλλουμε στους υπόλοιπους τις ευρωπαϊκές αξίες και να περιορίσουμε εκείνους τους γίγαντες των δεδομένων που έχουν ήδη δηλαδή στην κατοχή τους τεράστιους όγκους δεδομένων και τους εκμεταλλεύονται ε, να τους, να τους περιορίσουμε και να θέσουμε εμείς ε, τους όρους μας. Υπήρξαν για παράδειγμα ανταγωνιστές του Facebook οι οποίοι δεν κατάφεραν να ορθοποδήσουν λόγω των δικών μας περιορισμών ε, σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα ήθελα την άποψή σας ε, επ' αυτού. Διάβασα Κάτι ακόμη. Διάβασα ένα άρθρο στο Spiegel για το πόσο εύκολο είναι μέσω των, των, ε, δικτύων, ε, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να επηρεάσει κανείς την, ε, την κοινή γνώμη. Πώς μπορεί δηλαδή κάποιος από αντιδημοφιλής να γίνει μέχρι και πρόεδρος των, των ΙΠΑ. Πώς λειτουργεί λοιπόν αυτή η χειραγώγηση ε, μέσω των, στην ψηφιακή σφαίρα και πώς μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε. Αυτή θα ήθελα την, την άποψή σας από αυτού. κυρία Τσίπρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ε, συμφωνήσω με την προλαλή ε, και να πω και εγώ ότι και εγώ ε, δυσκολεύομαι λίγο με αυτά τα ψηφιακά θεμελιώδη δικαιώματα, γιατί έχουμε θεμελιώδη δικαιώματα και βλέποντας το κείμενό σας υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ήδη εξασφαλίζονται μέχρι του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είτε έρχομαι σε επαφή με κάποιον άνθρωπο, είτε έρχομαι σε επαφή μαζί του εικονικά, ε, η αξιοπρέπεια του, του καθενός είναι εξασφαλισμένη. Το ίδιο ισχύει και για το άσυλο της κατοικίας. Φυσικά σε αυτό συμπερι, συμπεριλαμβάνεται ε, ότι δεν θα επιτρέπεται για παράδειγμα δεν επιτρέπεται για παράδειγμα να υπάρχουν drones έξω από το σπίτι μου και να με παρακολουθούν. Γι' αυτό και ε, πιστεύω ότι αυτό που είπατε κύριε Σούλτς ότι είναι σωστό, ότι πρέπει να ελέγξουμε και να εξετάσουμε αν ε, υπάρχουν νέες προκλήσεις στην ψηφιακή σφαίρα και να δούμε αν πράγματι χρειάζεται να ρυθμίσουμε και νομοθετικά τα ζητήματα. Γιατί και η τάξη μεγέθους στο ψηφιακό κόσμο είναι διαφορετική από ότι στον αναλογικό κόσμο. Το... Να σας δώσω ένα παράδειγμα σε, ας πούμε ότι υπάρχει ένα bullying ενός ε, μαθητή από συμμαθητές του. Αυτό είναι ήδη άσχημο, όμως μεγεθύνεται αφάνταστα στον ψηφιακό κόσμο, γιατί εκεί μπορούν ξαφνικά να αρχίσουν να συμμετέχουν σε αυτό το bullying και σε αυτή τη διαδικασία άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ποτέ δει τα παιδιά αυτά όλα αυτά είναι πραγματικά πολύ σημαντικά ζητήματα και εκεί δεν θα χρειαστούμε μόνο, δεν θα, δεν θα αρκεί να, υπάρχουν νομοθετικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες. Θα χρειαστούμε και έναν κοινωνικό διάλογο, όπως αυτός, ο οποίος, αυτό, αυτός τον οποίο εσείς διοργανώσατε, για να δούμε πώς η κοινωνία θέλει να χειριστεί τις ψηφιακές δυνατότητες και τι προκλήσεις και τα προβλήματα. Και κάτι τελευταίο. Προστασία της ιδιωτικής σφαίρας. Το γεγονό ότι ο συνδυασμό διαφόρων δεδομένων τα οποία ε, δημιουργώ ε, σε διάφορες φάσεις της ζωής μου, κατά την αποστολή email, κατά τα ψώνια μου, κατά τη χρήση διαφόρων εφαρμογών, οδηγεί στο, στο ότι υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ποιος είμαι, ξέρουν τι μου αρέσει, τι κάνω, που ενδεχομένως ε, μπορούν να, να με εμπλέξουν ακόμη και σε ποινικέ διαδικασίες λόγω αυτών των γνώσεων που έχουν ε, επί του ατόμου μου. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν και νομίζω ότι και στο δικό σας κείμενο ε, περιλαμβάνεται και μια τέτοια ενότητα ότι χρειάζεται δηλαδή να ρυθμίζεται το, το, ο όγκος των δεδομένων που επιτρέπεται να γίνεται αντικείμενο χρήσης από άλλους, ε, πρέπει να περιοριστεί ο, δεδο... όγκος των δεδομένων ε, που μπορεί κανείς να αποθηκεύει για σένα. Χάρτα νομίζω ότι δεν χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε όμως σε κάθε περίπτωση μια συζήτηση για το ποιες καταχρήσεις και ποιοι κίνδυνοι μπορούν να ε, προκύψουν στην πορεία αυτής της ψηφιακής εποχής και όλα αυτά βεβαίως πρέπει να συζητηθούν σε βάθος. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία στοιχεία τα οποία τα θεωρώ σημαντικά στη διαδικασία. Ανήκω σε αυτούς που συζήτησαν το θέμα στην ομάδα, στην ομάδα των συντακτών του κειμένου. Είναι μια πρόταση για συζητήσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Χρειάζεται εμβάθυνση το ζήτημα. Να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να εφαρμόσουμε τα ισχύοντα θεμελιώδη δικαιώματα στον ψηφιακό κόσμο καλύτερα και πώς μπορούμε να τα διαβρύνουμε τα δικαιώματα αυτά μέσω συμπροματικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή συμπροματικών επεξηγήσεων όσον αφορά τα ισχύοντα ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα, ούτω ώστε να έχουμε ένα καλύτερο εφαρμοστέο πλαίσιο για την ψηφιακή εποχή. Χρειάζεται αυτή η συζήτηση, είναι απαραίτητη, πρέπει να γίνει και στο Ευρωκοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Ήταν γερμανική πρωτοβουλία αλλά θα πρέπει τώρα να μεταδοθεί αυτή η συζήτηση και σε άλλα βήματα ανοιχτών συζητήσεων στην Ευρώπη. Βέβαια δεν θα γίνει μια ανοιχτή η αλλαγή και η προσαρμογή αναγκαία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή της βασικής νομοθεσίας για να προσαρμοστούμε στην ψηφιακή πραγματικότητα. Ίσως στην επόμενη συνέλευση για τις συνθήκες σε 5-10 χρόνια να το καταφέρουμε. Αυτοί που θα ασχοληθούν με τις αλλαγές τότε θα πρέπει να λάβουν υπόψη την ιδέα προσαρμογής των θεμελιωδών δικαιωμάτων ώστε να καλύπτεται και η ψηφιακή εποχή. Άρα διεύρυνση και συμπλήρωση των δικαιωμάτων για το ψηφιακό περιβάλλον. Κάτι εξίσου σημαντικό. Θα ήταν υπέροχο να προωθηθεί αυτό ως πρωτοβουλία. Μόνο με ένα κείμενο στο τραπέζι μπορούμε να έχουμε μια βάση για συζητήσεις για να διαλυθούν οι νεφελώδεις προκλήσεις που αντιμετωπίσουμε. Χρειάζεται να είμαστε πιο λεπτομέρειες, πιο συγκεκριμένοι, αντί να ανταλλάσσουμε ορολογίες, που πολύ συχνά αυτό παρατηρείται στον ψηφιακό κόσμο. Η Βάρμπαρα Σπινέλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε Σούλτς. Ευχαριστώ καθηγητά Μπόντα. Χαίρομαι που η Χάρτα Θεμελιωδών ε, Δικαιωμάτων προτείνεται. Πιστεύω ότι είναι κάτι απαραίτητο. Ο διαδικτυακός κόσμος παρουσιάζεται σαν ένα κοινό αγαθό, κάτι που συνεπάγεται νέα είδη δικαιωμάτων ανωνυμία, δικαίωμα κύρωσης, να διαγράφονται τα στοιχεία, ψηφιακά, πνευματικά δικαιώματα κλπ. Διαβάζοντας τη χάρτα αυτή, τη δική σας, δοκίμασα να τη συγκρίνω με παρόμοια χαρτά. Ο καθηγητής Μπόντε τη γνωρίζει σίγουρα. Η διακήρυξη των δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, κάτι που ενέκρινε το Ιταλικό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2015. Κάνοντας τη σύγκριση των δύο αυτών κειμένων και θα έλεγα ότι η δική σας είναι άκρως ενδιαφέρουσα, με οδηγεί να υπογραμμίσω κάποια σημεία. Ίσως να σας ενδιαφέρουν να τα συμπεριλάβετε στη δική σας χάρτα. Στο προήμιο λοιπόν γίνεται λόγος για προκλήσεις και απειλές. Εγώ όπως και εσείς κύριε καθηγητά, κύριε Μπούντα, εγώ θα μιλούσα και για μεγάλες ευκαιρίες που δημιουργούνται και ανοίγονται με αυτό το μέσο. Δεν θα υπογράμμιζα ίσως τόσο πολύ τις απειλές, αλλά θα τις έθετα στο διατακτικό, εκεί στο σημείο του τι πρέπει να γίνει όταν υπάρχει παραβίαση της αξιοπρέπειας και τι γίνεται με την κατάχρηση της ελευθερίας της έκφρασης. Όσον αφορά τα άθρα 3 και 15, εν γέννη, το θέμα του ψηφιακού χάσματος, του digital divide, εγώ θα υπογράμμιζα τα κοινωνικά δικαιώματα και τη δυσκολία να προσαρμοστούμε στον ψηφιακό κόσμο. Δυσκολίες που έχουν κάποιες περιοχές να προσαρμοστούν στον ψηφιακό κόσμο, κυρίως ύπεθρος, ηλικιωμένοι άνθρωποι και άνθρωποι που κοινωνικά έχουν πρόβλημα να έχουν πρόσβαση με την ίδια ευκολία στον ψηφιακό κόσμο. Για το άρθρο 4. Αυτό αφορά την ασφάλεια. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ότι οι δυνάμεις της τάξης δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα ιδιωτικά στοιχεία. Και εξαιρέσεις θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εγγύησεω με βάση νομική για τη διαφύλαξη σημαντικών νομικών αρχών. Εγώ εκεί ίσως θα προσέθετα ότι οι εξαιρέσει είναι εφικτές μόνο με μια αιτιολογημένη άδεια δικαστικής αρχής. Αυτό το πήρα από την Ιταλική χάρτα που συνέταξε ο καθηγητής Ροντότα. Για το άρθρο 6 και το άρθρο 7 που εν γέννη ασχολούνται με το profiling και τον αλγόριθμο είναι σωστό, πολύ σωστό να πούμε ότι επιτρέπεται το profiling μόνο βάσει νομοθεσίας. Εγώ θα έλεγα ότι το profiling μπορεί να αποτελέσει δικείμενο ε, αντίρρησης από πλευράς των ανθρώπων, να υποβάλουν έσταση κατά αυτού. Είναι το δικαίωμα της ταυτότητας. Άρθρο 5. Data Protection και Data Sovereignty. Τονίζεται ότι χρειάζεται η συνένεση του χρήστη. όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων. Αυτό που προβλέπεται στην Ιταλική χάρτα που είναι σημαντικό είναι ότι αυτή η συνένεση μπορεί να ανακληθεί. Η συνένεση δεν είναι μόνιμη. Μπορεί να ανακληθεί. Και ένα ενδιαφέρον κείμενο από την Ιταλική χάρτα. Όμως, παρόλα αυτά, η συνένεση δεν μπορεί να αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία το τελευταίο σημείο, διακόπτει ο Πρόεδρος, όταν υπάρχει σημαντική ανισορροπία εξουσιών μεταξύ των ενδιαφερομένων ανθρώπων και εκείνων των εμπλεκομένων ανθρώπων, των αντικειμένων της έρευνας και εκείνων που διεξάγουν την έρευνα. Είχα και άλλα πολλά να πω, αλλά σας ευχαριστώ που με αφήσατε από αυτά. Μπάρμπαρα. Το, το διάβασες. Το διάβασες. Ε. Και ίσως ε, θα μπορούσε να συνεχίσει το διάλογο με τον καθηγητή Μπούντε. Ο κύριος ε, Όλσεν. Ευχαριστώ. Χαιρετίζω αυτή την πρωτοβουλία γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι εκτός κοινοβουλίου αλλά και άνθρωποι του κοινοβουλίου να ε, συνέρχονται και να συζητούν ε, και να αλληλεπιδρούν και να συνδιαμορφώνουν αυτού του είδους συζητήσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω και μια έκκληση, ενδεχομένως να μπορούσε να μας δοθεί περισσότερος χρόνος για να γίνει ακόμα πιο δημιουργικός αυτός ο διάλογος. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία αυτή, γιατί και ε, στα... Ε, ε, στα συμπεράσματα της Επιτροπής μας είχαμε διεκδικήσει και ζητήσει κάτι ε, παρόμοιο και θεωρώ ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Και στην ε, χάρτα για των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, έχουμε και ορισμένες διατυπώσεις όπου βεβαίως κάποιες από αυτές είναι και απαρχαιωμένες γιατί πράγματι διάφορα θέματα δεν είχαν ανακύψει καν ακόμη. Πάντως, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει κάποιο επιχείρημα κατά του να οξύνουμε τη ματιά μας ε, ή ως Ευρωπαίοι να αποτελέσουμε και ένα μοντέλο για τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, είναι σημαντικό να συνδιαμορφωθούν ε, οι ψηφιακές δομές και ακούμε πολύ συχνά και από τους Αμερικανούς φίλους ότι ε, πολλές φορές τους ε, ενδιαφέρει ε, αυτή η δουλειά που κάναμε όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πολλές φορές είχαν εκφράσει τις αντιρρήσεις τους, αλλά τώρα που ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή, φαίνεται ότι πολλές φορές οι Αμερικάνοι δείχνουν το ενδιαφέρον τους για την διαδικασία αυτή. Δεν έχουμε να κάνουμε άλλωστε με αχαρτογράφητα είδατα πλέον τόσο πολύ όσο ίσως στο παρελθόν σκέφτομαι διάφορα θέματα. Το μάρκετινγκ, τις εξατομικευμένες προσφορές, το δικαίωμα επιλογής. Υπάρχει εδώ πράγματι ένας κίνδυνος στρέβλωση τη αγορά, της ίδιας της λειτουργία, της οικονομίας της αγοράς, γιατί η αγορά προϋποθέτει ότι ο καταναλωτής έχει την επιλογή να διαλέξει το προϊόν που του αρέσει. Αντιθέτως, ε, ε, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αν βρίσκομαι εγώ σε μια ψηφιακή φούσκα και δεν γνωρίζω καν ποιε είναι οι δυνατότητε ή οι επιλογέ που έχω ε, μπροστά μου. Όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα που πρέπει να συζητηθούν σε βάθος και Χαίρομαι πολύ που και η Μπάρμπαρα Σπινέλη ε, έφερε και αυτή την ιταλική διάσταση, αν θέλετε, στη συζήτηση, γιατί ε, παρότι ξεκίνησε η συζήτηση αυτή από τη Γερμανία, πιστεύω ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να προσλάβει έναν ευρωπαϊκό, πανευρωπαϊκό χαρακτήρα για να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες όλων των ε, λαών της Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά, σας ευχαριστώ για την ε, πρωτοβουλία σας αυτή. Σας ευχαριστούμε. Πολύ σωστά ε, είπατε ότι αυτή η συζήτηση δείχνει πόσο προσφυλής ε, είναι η υπόθεση αυτή στην Επιτροπή μας και πόσο ζωηρό ενδιαφέρον δείχνουμε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον καθηγητή Μπούντε για ένα πεντάλεπτο μόνο, για να μην μείνουμε πίσω στα υπόλοιπα σημεία της ημερήσιας διάταξης και μετά ο πρόεδρος Σούλτς ε, θα ολοκληρώσει με κάποια συμπεράσματα. Θέλω να τονίσω τρία-τέσσερα σημεία. Κυρία Χόλμαϊρ, δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα έγγραφο φόβου, αλλά ένα έγγραφο ελευθερίας, το οποίο θα αναγνωρίζει το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα big data σήμερα. Υπάρχουν και διάφορες άλλες δυνατότητες συνδυασμού ε, δεδομένων, τεχνικών και μη. Και γι' αυτό το λόγο ανακύπτουν νέα ερωτήματα που δεν αρκεί κανείς μόνο να έρθει και να νομοθετήσει, αλλά χρειάζεται πρώτα απ' όλα να τα κατανοήσει σε βάθος. Είναι πολύ σημαντικό για αυτό το νέο τομέα του δικαίου να υπάρξει μια κοινή αντίληψη και μια κοινή κατανόηση των ζητημάτων. Δεύτερον, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, προφανώς και δεν είναι ούτε μόνο γερμανικό το θέμα αυτό, ούτε καν ευρωπαϊκό και μόνο. Και γι' αυτό βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το ότι ε, θα μπορούσαν οι πρωτοβουλίες που υπάρχουν ήδη σε εθνικό επίπεδο να συνδυαστούν σε μια ενδεχομένως πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Αν σκεφτεί κανείς τα έξυπνα σπίτια και μόνο, κατανοεί κατευθείαν ότι η ίδια η ιδιωτικότητα μεταμορφώνεται και προσλαμβάνει έναν διαφορετικό χαρακτήρα εποχή. Χρειάζεται λοιπόν νέες προσεγγίσεις, νέες πρωτοβουλίες για το πώς θα εξασφαλίσουμε και θα εγγυηθούμε την ιδιωτικότητα στη νέα εποχή. Υπάρχει λοιπόν για μια νέα γενιά ότι, η, αντίληψη ότι το, το, δημόσιο ε, αγαθό μπορεί ταυτόχρονα να είναι και ιδιωτικό, ατομικής ιδιοκτησίας. Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένας νέος δημόσιος χώρος μέσα από συνδυασμό ατομικοτήτων. Και αυτό που αναφέρατε ως δημιουργία φούσκας ψηφιακής χρειάζεται να απαντηθεί και να συζητηθεί γιατί αποτελεί ένα βασικό ερώτημα και των νέων ταξικών δομών της κοινωνίας μας, οι φούσκες της, της ε, ψηφιακής σφαίρας. Τελευταίο ερώτημα που πρέπει να συζητηθεί, κυρία Ζήπλη το, θέσατε κι εσείς, μήπως τελικά τα δεδομένα αποτελούν μια, ε, μια νέα μορφή του δημόσιου αγαθού ποια είναι δημόσια αγαθά, ποια είναι ιδιωτικά αγαθά, ποια είναι αυτά τα δεδομένα και πώς θα τα ταξινομήσουμε. Όλα αυτά ε, απαιτούν να γίνει μια τεράστια συζήτηση και σε βάθο. Για την ανακεφαλαίωση Ξεκίνησα να εργάζομαι από αυτό το θέμα πριν από 22 χρόνια. Κοιτάζοντα λοιπόν την εξέλιξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων αυτά τα 22 χρόνια, στις συνθήκες και στα εθνικά συντάγματα που ισχύουν. Κυρία Ζίπελ και κύριοι ε, συνάδελφοι, ε, συμφωνώ μαζί σας, αλλά πριν από 22 χρόνια εγώ δεν θα μπορούσα να είχα φανταστεί ότι τα ατομικά δικαιώματα, ε, θέσατε αυτό το καταπληκτικό παράδειγμα του μαθητή που δέχεται bullying από τους μαθητές τους, ότι θα μπορούσαν ποτέ τα πράγματα να φτάσουν εδώ. Οι τεχνολογικές εξελίξεις λοιπόν είναι πολύ γρηγορότερες πολλές φορές από ό,τι μπορούμε εμείς ως νομοθέτες να παρακολουθούμε για να δημιουργούμε και τις κατάλληλες και τις ενδεδειγμένες ε, δομές. Για ποιο λόγο λοιπόν ξεκινήσαμε αυτή την πρωτοβουλία ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη μας έθεσε και το παράδειγμα των, ε, των ε, ανθρώπων που έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Αυτό που ε, ενδιαφέρει εμένα προσωπικά είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το ο φορέας και, και το όργανο που κυρώνει διεθνείς συμβάσεις. Άρα το ερώτημα για το πώς θα γίνει ο συνδυασμός του big data και του big commerce, για παράδειγμα, το αν θα παραβιάσει ή θα επηρεάσει τα ατομικά δικαιώματα γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος όταν τα δεδομένα των ε, ατόμων γίνονται αντικείμενο εμπορίας, οικονομικής εκμετάλλευσης, που δεν μπορεί πλέον να τα εγγυηθεί ε, το κράτος, αλλά αντιθέτως τα κράτη δεν μπορούν πια να εξασφαλίσουν τα ατομικά δικαιώματα τα δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ατόμων, ακριβώς γιατί ε, υπάρχει αυτή η ασυμμετρία σε σχέση με τις τεχνολογικές εξελίξεις που τρέχουν. Το γεγονός όμως ότι το αντιπροσωπευτικό σώμα, το σώμα των, των βουλευτών, αυτό που σταμάτησε τη συγκέντρωση δεδομένων στον, στον τραπεζικό τομέα και μόνο και ως εκ τούτου σταμάτησε και μια σχετική συμφωνία με τις ΗΠΑ, μας οδήγησε στο, ε, στη διαπίστωση και στο ερώτημα πού θα μπορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλει σε αυτή τη συζήτηση, πού θα μπορούσαν τα εθνικά ε, κοινοβούλια να συμβάλλουν σε αυτή τη συζήτηση. Φυσικά δεν είναι γερμανικό το θέμα, είναι μια παγκόσμια συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ευχαριστώ πολύ ακόμα και για τις κριτικέ σκέψεις που εκφράστηκαν. Για το αν χρειαζόμαστε μια τέτοιου είδου νέα χάρτα ψηφιακών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το είπα και εισαγωγικά κυρία Χόλμαϊρ. Εμείς δεν έχουμε έρθει εδώ για να ε, εγκρίνουμε μια νέα χάρτα. Ε, ούτε αυτό ήταν ο σκοπός της ομάδας μας. Ιδιώτε ως, ε, ενεργώντας ως ιδιώτες συνήλθαμε, συγκεντρωθήκαμε και συζητήσαμε αυτά τα ζητήματα για έναν περίπου χρόνο και μάλιστα διαφωνήσαμε και πολύ και ε, στο τέλος και ο κύριος Μπούντε αλλά και οι συνάδελφοι όπως ο Ζάς ε, Λόμπο ή ο Βάλτερ Σπίτς που συζητήσαμε αυτά τα θέματα συζητήσαμε, διαφωνήσαμε και στο τέλος καταλήξαμε και συμφωνήσουμε ότι πρόκειται για ένα προσχέδιο κειμένου. Γι' αυτό λοιπόν ε, χρειαζόμαστε ακόμη και την διαφωνία και την, τις προκλήσεις γιατί πρέπει να συζητηθεί το θέμα. Τα υπάρχοντα μέσα και εργαλεία επαρκούν για την εποχή. Εγώ προσωπικά πιστεύω όχι. Παρ' όλα αυτά, η όλη αυτή συζήτηση θα ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία που χρειαζόμαστε. Μια χωρίς αποκλίσεις και διακρίσεις συζήτηση σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και γι' αυτό ε, ευχαριστώ πολύ και το Ίδρυμα της εφημερίδας Zeit. Δεν θέλουμε αυτή η συζήτηση να περιοριστεί στους πολιτικούς αλλά να συμμετάσχουν σε αυτήν ενεργά και οι πολίτες. Στο τέλος της όλης διαδικασίας φυσικά το θέμα αυτό θα συζητηθεί στο κοινοβούλιο αλλά όχι σε όλη τη διαδικασία πρέπει να έχει προηγηθεί σε βάθος συζήτηση σε όλη την κοινωνία. Ο κύριος ε, συνάδελφος Χόλτσερ το είπε και έχει δίκιο. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Μα συμφωνώ απολύτω. Γι' αυτό και σα παραδίδουμε σήμερα αυτό το προσχέδιο κειμένου για να μπορέσετε με τον χρόνο σα να συζητήσετε και να το εξετάσετε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να, να τονίσω και κάτι ακόμη. Υπάρχουν εδώ, ε, σε αυτή την αίθουσα, συνάδελφοι που ε, με κατηγορούν στη διάρκεια της ε, θητείας μου ότι δεν είμαι αρκετά ευαίσθητος ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ένας από αυτούς τους συναδέλφους μάλιστα έλαβε και το λόγο εδώ στη συζήτηση. Και γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει λίγο δεν είμαι αυτό που θα έλεγε κανείς ο πάπας της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Το αντίθετο. Υπάρχουν συνάδελφοι που βρίσκονται ε, εδώ μέσα και που με έχουν κατηγορήσει ότι είμαι υπερβολικά ε, γενναιόδωρος ε, ή ενδεχομένως ακόμη και απρόσεκτο σε σχέση με, με αυτό το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτούς τους συναδέλφους θέλω να τους ευχαριστήσω. Γιατί στη διάρκεια των τελευταίων ετών, ιδίω κατά την κύρωση συμφωνιών, μου άνοιξαν τα μάτια για το πόσο πίσω έχουμε μείνει όσον αφορά την εξασφάλιση και την εγγύηση των ψηφιακών θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή. Και αν ο αναλογικός κόσμος υποχωρήσει όλο και περισσότερο, κάποια στιγμή ε, θα αρχίσουν να θολώνουν και τα σύνορα μεταξύ αναλογικού και ψηφιακού κόσμου και γι' αυτό θα χρειαστούμε και νέες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να, να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα ψηφιακά και μη. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι μου δώσατε κίνητρο και το έναυσμα για να ασχοληθώ με αυτά τα θέματα και για να συμμετάσχω ενεργά σε αυτή τη συζήτηση να ξαναπώ με αυτό που, ε, αυτό που είπε ο Γιώζεφ Βάιντενχόλτσα. Και μια παράκληση. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε στη Γερμανία, πράγματι. Αλλά επιθυμώ και εύχομαι να διευρυνθεί η συζήτηση αυτή και μέσω της συμβολής της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε Πρόεδρε Μάρτιν Σούλς και καθηγητά Μπούντε. Ε, αυτός είναι ο στόχος ε, και η επιθυμία και των συντονιστών να διευρύνουμε τη συζήτηση ώστε να λάβει ευρύτερο χαρακτήρα και ε, συμφωνούμε απόλυτα και υπάρχει απόλυτη σύμπνοια μεταξύ μας. Και όντως ε, έδειξε σε ζωηρό ενδιαφέρον ε, για όλα αυτά τα θέματα καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σου. Σας ευχαριστούμε θερμά και θα δώσουμε συνέχεια στο έργο που μας παρουσιάσατε σήμερα. Ευχαριστώ. Colleagues, we can um, Ωραία, συνάδελφοι, μπορούμε να περάσουμε μέσα στο επόμενο θέμα, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω. Σημείο 5. Όπως ξέρετε, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, έχουμε μια ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διακόπτω λίγο για να δώσω το χρόνο στο Ματία Σουρίτε, το Γενικό Διευθυντή, να λάβει θέση. Όπως είπα λοιπόν, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, έχουμε ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή συγκεκριμένων συμφωνιών επανεισδοχής. Ήρθε αυτή τη στιγμή και πάλι. Έχουμε δύο εκθέσεις ε, για τις ε, εκκρεμής εργασίε ό,τι αφορά τις διάφορες συμφωνίες επανεισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτων Χωρών και την, το σχέδιο κοινή πορείας σε θέματα μετανάστευσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Αφγανιστάν. Ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Ρούτε, θα μας κάνει την ενημέρωση γιατί δεσμεύτηκε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες τις τη συμφωνίες επανεισδοχής τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να μας ενημερώνει κάθε εξάμεινο για την εφαρμογή αυτών των συμφωνιών επανεισδοχής με ειδική μνήμα των τρέχουσών εργασιών για την των εργασιών της, των κοινών επιτροπών επανεισδοχής που παρακολουθούν και διευκολύνουν την εφαρμογή της συμφωνίας. Μάλιστα, 14 Νοεμβρίου, οι συντονιστές αποφάσισαν να θέσουν αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη, το θέμα του σχέδιου κοινής πορείας θέματα μετανάστευση με το Αφγανιστάν και γι' αυτό το συμπεριλάβαμε στη σημερινή ημερήσια διάταξη γιατί αφορά θέματα επανεισδοχή. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στο Γενικό Διευθυντή τον κύριο Ρίτε, καλώ ορίζοντα τον και του δίνω το λόγο. σα. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους σας. Και μετά τη συναρπαστική συζήτηση που είχατε για το ψηφιακό πρόγραμμα εργασιών και τα ψηφιακά θεμελιώδη δικαιώματα, εγώ ναι, νιώθω ότι περισσότερο ενημέρωση κάνω και όπως σωστά είπατε κύριε Πρόεδρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει την υποχρέωση να σας ενημερώνει άπαξ το εξάμεινο ε, για τις συμφωνίες επανειστοχής ε, που έχουμε συνάψει και μάλιστα την τελευταία φορά που είχα έρθει εδώ ήταν το Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά. Οπότε πέρασε πάλι ένα εξάμεινο και ήρθε η ώρα να σας ε, κάνω μια νέα ενημέρωση. Θα ήθελα πρώτα να πω λίγα λόγια γενικά. Ο επαναπατρισμός των παράτυπων μεταναστών αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα μιας ε, βιώσιμης διαχείρισης της μετανάστευσης. Και μάλιστα οι παράτυποι μετανάστες ε, ε, θα έχουν λιγότερε πιθανότητε να χάσουν τι οικονομίε τη χώρα των, των οικογένειών του, των κοινοτήτων του και να διακινδυνεύουν σε επικίνδυνα ταξίδια, να παίζουν κοροναγράμματα τη ζωή του αν συστηματικά επαναπατρίζονται στη χώρα προέλευση του. Θα διακινδύνευαν πολύ λιγότερο. Γνωρίζετε τα νούμερα. Σήμερα έχουμε μόνο 40% περίπου του συνόλου των αποφάσεων επιστροφής ε, που δυστυχώς ε, μόνο το 40% εφαρμόστηκε από τις αποφάσεις αυτές επιστροφής και οι περισσότεροι, παρόλο που έχουν δει τις αιτήσει του ασύλου να απορρίπτονται, έχουν καταφέρει να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα πολύ συχνά σε επισφαλείς συνθήκε. Κάτι που μας επαναφέρει στη γνωστή συζήτηση για τη σωματοεμπορία, το δουλεμπόριο, την χρήση ε, ξαναγκαστικής εργασίας και ούτω καθεξής. Σε ό,τι αφορά τώρα τις πολιτικές επαναπατρισμού επιστροφής, αυτές προσκρούν σε πολλά αριθμά εμπόδια. Καταρχήν, έχουμε κάποιες περιπτώσεις όπου νομοθεσία που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους χρήζοντες στη διεθνή προστασία, ε, τέτοια νομοθετήματα να τη χάνουν κατάχρησης. Επίσης έχουμε νομοθετικές διατάξεις και διοικητικές πρακτικές στα κρατη που επηρεάζουν συστήματα ασύλου και επιστροφής που επιβραδύνονται πρώτη, για διαδικασίες που επιβραδύνονται, που εμποδίζουν την επιστροφή και πολλές φορές αυτή η έλλειψη επιστροφής οφείλεται σε έλλειψη συντονισμού μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των κρατών μελών, των αρμοδίων υπηρεσιών μετανάστευσης ή επίσης οι υπηρεσίες ασύλου δεν έχουν αρκετές ικανότητες, ανεπαρκή κέντρα υποδοχής, ανεπαρκή κέντρα κράτησης και το καθεξής. Αυτά ως προς τις αδυναμίε που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλο μείζον εμπόδιο όμω είναι και αυτή ε, η πρακτική της, ε, του επαναπατρισμού ε, μεταναστών χωρίς έγγραφα. Γιατί πολύ συχνά έχουμε μετανάστες που είτε χάνουν τυχαία είτε καταστρέφουν σκεμένα τις ταυτότητές τους, τα διαβατήριά τους. Έχουμε παράτυπους μετανάστες που αρνούνται να συνεργαστούν με τις αρμόδιες αρχές Οπότε χρειαζόμαστε την ε, πλήρη συνεργασία με τη χώρα προέλευσης αυτών των ε, ανθρώπων. Με, προκειμένου να έχουμε ε, αναγνώριση και επανέκδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων. Κάτι που προϋποθέτει αγαστή συνεργασία, ταχεία συνεργασία και με προξενία, με προξενικές αρχές, αλλά και με τις εθνικές αρχές των τρίτων χωρών. Θα ήθελα τώρα να σας δώσω μερικά παραδείγματα δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε σε θέματα συνεργασίας. Με βάση το Διεθνές Τελωνιακό Δίκαιο, κάθε χώρα έχει υποχρέωση να επιτρέψει στους υπηκόους, ε, τους, στους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Μερικές φορές όμως έχουμε περιπτώσεις που οι χώρες αρνούνται να εκδώσουν ταξιδιωτικά έγγραφα στους υπηκόους τους. Είτε χρονοτριβούν, είτε εκδίδουν ε, πολύ καθυστερημένα όταν πια έχουμε χάσει τα ίχνη των παράτυπων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή έχουμε χώρες που αρνούνται να δεχθούν ε, επαναπατρισμό των υπηκών τους με συγκεκριμένες τσάρτερ πτήσεις. Μερικές φορές έχουμε ζητήσει να έχουν ζητήσει να γίνονται επιστροφές μόνο με τις εθνικές αερογραμμές. Επίσης έχουμε προξενία που μερικές φορές ε, δίνουν συμβουλές στους υπηκόους τους ε, ε, πώς να χρονοτριβήσουν, πώς να κολλησιεργούν ώστε να παρατείνουν την παραμονή τους στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Και γι' αυτό στις διαπραγματεύσεις που έχουμε με τρίτες χώρες προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ κινήτρων και αντικινήτρων σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη αλλά και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων ώστε να δημιουργήσουμε ένα περιεκτικό πλαίσιο συντονισμού. Και το 2016 καταφέραμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό και να υιοθετήσουμε μια πιο συστηματική και συγκροτημένη προσέγγιση ε, ώστε να βελτιστοποιήσουμε την επιρροή μας στις τρίτες χώρες και να ε, βελτιστοποιήσουμε επίσης ε, την επιρροή και την συνάφεια μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών μας. Ε, μερικές φορές όταν με ακούω, <laughs> ακούω τα λόγια μου, λέω, Μήπω είναι κανένα άκαρδο αυτός ο άνθρωπο. Τι άκαρδο τι ανέστητο που είναι. Όχι. Μην με παρεξηγείτε. Εδώ μιλούμε για ανθρώπου ε, που πέρασαν από τη διαδικασία, έκαναν, υποβίβαλαν αίτηση και του αρνήθηκε, ε, απορρίθηκε το αίτημα χορήγηση ε, διεθνού προστασία, έχουν εξαντλήσει τι νόμιμε διαδικασίε και εμπίπτουν στην διαδικασία επιστροφής. Είναι επιλέξιμη για επιστροφή. Γιατί πολύ συχνά γίνεται σύγχυση μεταξύ των προσφύγων αφενός και των παρατύπων μεταναστών αφετέρου. Εδώ μιλούμε για παράτυπους μετανάστες και η προσέγγιση που εθετήσαμε φέτος έχει αποφέρει καρπούς και σε συνεργασία με τις τρίτες χώρες έχουμε περιορίσει το, τη σωματιμπορία και την λαθροδιακίνηση. Αλλά για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, οφείλω να ομολογήσω ότι τα νούμερα δεν έχουν αλλάξει. Πάλι είμαστε γύρω στο 40% της εφαρμογής των ηλυμένων αποφάσεων επιστροφής. Οπότε από αυτή την άποψη η νέα μας προσέγγιση δεν έχουν δείξει μετρήσιμα αποτελέσματα τουλάχιστον. Γι' αυτό και η επανεισδοχή έχει αναχθεί σε μείζωνα προτεραιότητά μας ε, σε όλες τις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες. Και θα ήθελα να τονίσω ότι δεν μιλούμε εδώ για σύναψη μια συμφωνίας, υπογραφή μιας συμφωνίας επανεισδοχής ε, καθ' αυτή, αλλά μιλούμε για συγκεκριμένη βελτιωμένη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης. Αυτή είναι πολύ πιο σημαντική από μια μηγή υπογραφή συμφωνίας επανεισδοχή. Αυτές είναι οι αδρές γραμμές και το πλαίσιο των διαφόρων ε, συμφωνιών επανεισδοχής. 17 είναι οι συγκεκριμένες ε, συμφωνίες επανεισδοχής. Δεν πρόκειται να τις αναλύσω διεξοδικά γιατί θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Εν συντομία θα σας κάνω μια παρουσίαση ξεκινώντας από την Τουρκία. Η συνεργασία με την Τουρκία για την επιστροφή και επανεισδοχή ε, διευρύνθηκε δεόντως με την δήλωση της 18ης ε, Μαρτίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Και μάλιστα με τη ε, διακήρυξη αυτή θελήσαμε να εξαρθρώσουμε τα μοντέλα, επιχειρησιακά μοντέλα των λαθροδιακινητών που εκμεταλλεύονται τους ε, μετανάστες και να προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τη παράτυπη ροή μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα και να αποτρέψουμε ανθρώπινες τραγωδίες ε, αγνοωμένων ή ε, ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους, ε, που θαλασσοπνίγονται, που χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Και μάλιστα από τη κοινή διακήρυξη με την Τουρκία έχουμε δυστυχώς καταγράψει περίπου 63 νεκρούς και αγνοωμένους στο Αιγαίο. Την ίδια περίοδο βέβαια, το 2015, είχαμε πάνω από 490 θανάτους ανθρώπων που πνίγηκαν δηλαδή, έχασαν τη ζωή τους, προσπάθησαν να διαπλέψουν ε, τη μικρή αυτή απόσταση από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά. Την Τετάρτη μάλιστα δημοσιεύσαμε και την έκθεσή μας, την τέταρτη έκθεση που παρουσιάζει διεξοδικά την πρόοδο που σημειώσαμε ως προς την κοινή διακήρυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας και απαριθμούμε και τις δεσμεύσεις και το βαθμό εκτέλεση αυτών των δεσμεύσεων αυτής της διακήρυξης. Σε ό,τι αφορά την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών από τα νησιά, μέχρι στιγμής η Τουρκία έχει δείξει έγκαιρη και αγαστή διάθεση συνεργασίας και παρά τις ε, δυσκολίες που είχαμε το καλοκαίρι μετά την ε, απόπειρα πραξικοπήματος, έχουμε μέχρι στιγμής 1.187 ε, παράτυπους μετανάστες που έχουν επιστρέψει με βάση το διμερές πρωτόπολο Ελλάδος-Τουρκίας στα πλαίσια της διακήρυξης και με βάση το σύστημα ε, το σύστημα 1 προς 1, 2.426 Σύριοι έχουν επανακατασταθεί από την Τουρκία σε διάφορα κράτη-μέλη και περιμένουμε ακόμη 230 να μετακατασταθούν μέχρι τα τέλη του έτους. Είναι αλήθεια ότι ο αριθμός των επιστροφών από τα νησιά προς την Τουρκία εξακολουθεί να παραμένει χαμηλός εξαιτία του αργού ρυθμού της επεξεργασίας του υψηλού αριθμού αιτήσεων ασύλου. Οι ελληνικές υπηρεσίες ε, έχει διπλασιάσει τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων που απασχολούνται στα νησιά για τη διεκπαιρέωση αυτών των αιτήσεων και μάλιστα θα προσληθούν και άλλοι εμπειρογνώμονες μέχρι τα τέλη του έτους. Η Συμφωνία Ευρωπαϊ... Ε, Παρισδοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ε, θα πρέπει να θεωρηθεί και υπό το πλαίσιο των συζητήσεων για την, την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Έγινε κάποια πρόοδος ό,τι αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας Επανεισδοχής το 2016. Είχαμε δύο ε, κοινέ επιτροπέ επανεισδοχή και δύο τεχνικέ συνεδριάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εκπροσώπου των κρατών μελών και των τουρκικών αρχών και σε αυτές τις επιτροπές συζητήσαμε τις λεπτομέρειες των ε, εμποδίων ε, που συναντούμε στην εφαρμογή αυτής της ε, συμφωνίας επαρισδοχής. Η υποχρέωση επαρισδοχής Τούρκων υπηκών και οι σχετικές διατάξεις ισχύουν από το 2014. Η αριθμή βέβαια δεν είναι και πολύ εντυπωσιακή. Είναι χαμηλή, κάτω από 376 έχουμε και μάλιστα οι μισές αιτήσει έχουν γίνει δεκτές από την Τουρκία. Και λιγότερο από το 1 τρίτο των ε, Τούρκων υπηκών έχουν πραγματικά επιστραφεί. Περίπου 100. Και αυτά είναι τα στοιχεία του 2016 που προηγούνται της απόπειρας πραξικοπήματος. Εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στη συνεργασία μας με τα προξενία, με τις προξενικές αρχές. Πάντως, γενικώ η συνεργασία με την Τουρκία έχει βελτιωθεί. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βέβαια δεν εφαρμόζει τις διατάξεις για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Συμφώνησε βέβαια ότι θα σημειώσουμε κάποιο πρόοδο, αυτό το έχει υποσχεθεί στην προηγούμενη συζήτηση για την απελευθέρωση των θεωρήσεων, αλλά η νομική οριστικοποίηση, τουλάχιστον αυτή είναι η ερμηνεία που υιοθετεί η Τουρκία, για να προχωρήσουν οι συμφωνίες επανειστοχής, ώστε να καλύπτουν και τους υπηκόους τρίτων χωρών, ε, με την ερμηνεία που δίνει η Τουρκία συνδέει αυτό το θέμα της κάλυψης και των υπηκών τρίτων χωρών με το ζήτημα της απελευθέρωση των θεωρήσεων. Πάντως συνεχίζουμε τον επικοδομητικό διάλογο μας με την Τουρκία και σας διαβεβαιώ, όπως έκανε και ο Επίτροπος Αβραμόπουλος και ο Αντιπρόεδρος μας και άλλοι, ότι το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων για την Τουρκία θα προταθεί μόνο μετά την υλοποίηση όλων των συγκριτικών κανόνων. Τώρα για την Τουρκία ένα άλλο στοιχείο που είναι σημαντικό αφορά τη Βουλγαρία. Η Τουρκία έχει διμερή συμφωνία και με την Βουλγαρία και βάσει αυτής έχει αναλάβει τη δέσμευση να βρει κάποιες ε, ε, πρακτικές λύσεις σε συνεργασία με τη Βουλγαρία. Κάτι που όμως δεν έχει γίνει ακόμη. Δεν έχουν βρεθεί ακόμη ικανοποιητικές ρυθμίσεις μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας. Αυτά ως προς την Τουρκία. Πάμε στο Πακιστάν. Το Πακιστάν είναι σημαντική χώρα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για επανεισδοχή. Να σας δώσω κάποια στοιχεία. Το 2015 είχαμε δραματική αύξηση Πακιστανών που έφταναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αύξηση 1000%. Είχαμε 43.000 ανθρώπους από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο. Άλλους 8.000 Πακιστανούς παράτυπους μετανάστες που δήλθαν τα σύνορα. Η συμφωνία επανεισδοχής που έχουμε το Πακιστάν, που ισχύει από το 2010, βοήθησε το 2014 να αυξήσουμε τον αριθμό των επιστροφών κατά 52, στο 52% αλλά μέχρι το του 2015 έπεσε το ποσοστό επιστροφών στο 36% περίπου και είχαμε και πολλές αρνητικές δηλώσεις που είχε κάνει ο Υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν συνέτεινε αυτό. Πήγε ο Επίτροπο Αβραμόπουλο τον Νοέμβριο του 2015 στο Πακιστάν και είχαμε δύο κοινέ επιτροπέ, συνεδριάσει τη Επιτροπή αυτή τη Ευρωπαϊκή του Πακιστάν, Φεβρουάριο και τον Ιούλιο. Έγιναν συνεδριάσει. Υπάρχουν πολιτικά εμπόδια ε, τα οποία ξεπεράστηκαν για την εφαρμογή τη συμφωνία, αλλά η γενική εικόνα πόρα απέχει το τέλειον. Κάποια κράτη-μέλη αναφέρουν ότι υπάρχει καλή συνεργασία, άλλες ότι έχει βελτιωθεί η συνεργασία, άλλες χώρες εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για συνεχείς πρακτικές ε, δυσκολίες. Τους τελευταίους μήνες είχαμε μια θετική εμπειρία με κοινέ επιχειρήσεις επιστροφών υπό το συντονισμό της Frontex με τη συμμετοχή κάποιων ευρωπαϊκών χωρών, μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από την άλλη έχουμε και περιπτώσεις όπου τα κράτη-μέλη υπέβαλαν αιτήματα επανεισδοχής χωρίς να λάβουν απάντηση από την πακιστανική πλευρά. Προσπαθούμε να υπάρχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα όσον αφορά τις σχέσεις μας με το Πακιστάν και θα το θέσουμε το ζήτημα στην επόμενη συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής επανιστοχής τον Ιανουάριο στις Βρυξέλλες. Τρίτη μεγάλη ομάδα, ανατολική εταιρική σχέση, ε, η Ρωσία, Δυτικά Βαλκάνια. Η ελοποίηση η εφαρμογή των συμφωνίων επανιστοχής με αυτές τις χώρες είναι αρκετά ικανοποιητική, πολύ ικανοποιητική θα έλεγα. Σταθερά τα ποσοστά, υψηλά ποσοστά επανιστοχής 81% Ουκρανία, 76% Μολδαβία, 67% Ρωσία, έγινε 16η συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε τον Ιούλιο επιβεβαίωσε την καλή εφαρμογή της Συμφωνίας Επανιστοχής και τώρα ξεκινάμε τη συζήτηση για την χρήση ηλεκτρονικών διάβλων ε, για τη διαβίβαση ετοιμάτων επανιστοχής σε επαφή με τις ρωσικές αρχές θα εφαρμόσουμε πιλωτικό πρόγραμμα μέσω βιντεοδιασκέψεων. Τρία κράτη-μέλη θα συμμετάσχουν. Η συνεργασία εν γέννη είναι καλή. Προφανώς βέβαια υπάρχουν κάποια πολιτικά στοιχεία που παρισφρίουν από καιρούς καιρών, διαβατήρια Φερρυπίν, που εκδίδονται στην Κρυμαία, που έχουν εκδοθεί στην Κρυμαία, για να σας δείξω ότι δεν είναι πάντα εύκολες αυτές οι σχέσεις. Όσον αφορά τη γεωργία, πολύ αποτελεσματική είναι η συνεργασία. Υπάρχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών. Τη χρησιμοποιεί ο φορέας IOM. Έχει γίνει ένα πρότυπο όσον αφορά τη διαχείριση των διαφόρων υποθέσεων και τις αιτήσει επανεισδοχής. Αρμενία, Αζερβαϊτζάν. Θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα εκεί, αλλά έχουμε βελτίωση. Η Αρμενία δεν είναι σε πιο μειονεκτική θέση από το Αζερβαϊτζάν και η εφαρμογή τη συμφωνής επανεισδοχής με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι πολύ ικανοποιητική. Ποσοστά επιστροφών που ξεπερνούν το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως του 42%, Αλβανία 87% και λοιπά και ούτω καθεξής. Τέλος, κάτι εξίσου σημαντικό. Πράσινο ακροατήριο. Καπ ε, Είναι η μόνη Αφρικανική χώρα με την οποία έχουμε και εφαρμόζουμε συμφωνία επανεισδοχής. Πάνε καλά τα πράγματα. Ξέρω ότι θέλετε να μας σταματήσετε, Πρόεδρε. Δεν θα πω κάτι για τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις, για τις συμφωνίες επανεισδοχής. Ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις με τέσσερις χώρες, αυτό να πω μόνο. Μαρόκο, Λευκορωσία, την και Νιγηρία. Συνεχίζονται αυτές. Μάλιστα αρκετές από τις διαπραγματεύσεις είναι μακροχρόνιες και τρεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα επίσημα, Ιορδανία, Αλγερία και Κίνα. Για διάφορους λόγους δεν έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσει. Αυτά για να σα δώσω μια γενική εικόνα του θέματος των επανεισδοχών. Ίσως θα θέλατε να υποβάλλετε ερωτήσεις και μετά να απαντήσω σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ κύριε Ρέιτε. Έχουν μεγάλη εμπειρία τα μέλη μας για το θέμα και θα έχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μέχρι 16.45 έχουμε στη διάθεσή μας. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και με το χρόνο, γιατί είναι η μοναδική ευκαιρία που έχουμε την δυνατότητα να λάβουμε πληροφορίες το σοβαρότερο το θέμα των επανεισδοχών. Ένα-δύο λεπτά ο καθένα παρακαλώ και ακριβώς το ψητό τη ερώτησή σας για να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά θα έχουμε και τον Υπουργό που θα έρθει στις 16.45. Η κυρία Σίπελ, ακολουθώ τη σειρά με την οποία ζητήσατε το λόγο. Έχει πάνω από δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με κάποιες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Μπορείτε να μας πείτε για μια ακόμη φορά γιατί το Κοινοβούλιο δεν αναμειγνύεται στην ε, διαμόρφωση αυτών των συμφωνιών επανεισδοχής. Δεύτερη ερώτηση, γιατί οι συμφωνίες επανεισδοχής δεν αποκαλούνται τούτο τρόπο. Αναφέρομαι στη συμφωνία με την Τουρκία και την κοινή προσέγγιση, την κοινή πορεία. δεν αναφέρεται σαν συμφωνία επανεισδοχής, έχει άλλο τίτλο. Τρίτον, όταν μιλάτε για επανεισδοχή, μπορείτε να μας πείτε κάτι έτσι γενικό. Αναφέρεται στους πολίτες της συγκεκριμένης χώρας ή και σε υπηκόους τρίτων χωρών. Αν σε όλες τις περιπτώσεις αναφέρεται σε υπηκόους τρίτων χωρών, γιατί στο καλό τόσο φτωχέ χώρες να παίρνουν υπηκόους τρίτων χωρών και εμείς να μην μπορούμε να τους φροντίσουμε. Κάτι άλλο που αναφέρατε, μια κοινή προσέγγιση για την επανεισδοχή, περιγράψατε κάποιες δυσκολίες στον τομέα αυτό για μια κοινή προσέγγιση για την επανεισδοχή. Δεν πρέπει καταρχάς να γίνει περισσότερη δουλειά για να έχουμε μια κοινή προσέγγιση για το πώς αποφασίζουμε αν σε κάποιον θα χορηγηθεί καθεστώς ασύλου ή όχι. Διότι διαφέρουν κατά πολύ οι αριθμοί από χώρα σε χώρα, από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Τελευταία ερώτηση. Ακόμα και αν κάποιος δεν τύχει ασύλου Ίσως να υπάρχει ανθρωπιστικός λόγος για να αφήσουμε τον άνθρωπο αυτό να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε κοινή προσέγγιση σε όλα τα κράτη-μέλη ή έχουμε και εδώ μεγάλες διαφορές. Και τι σημαίνει κάτι τέτοιο για την επανεισδοχή. Α, και κάτι τελευταίο. Κίνα. Πόσους πρόσφυγες έχουμε ερχόμενους από την Κίνα. Η κυρία Χόλμαν έρχεται το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά το ερώτημα τι συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους που επαναπατρίζονται στο Πακιστάν, για παράδειγμα, όπου επικρατούν πολύ δύσκολες συνθήκες, ακόμη και συγκρούσεις εχθροπραξίες. Μπορείτε να μας εξηγήσετε ποια μέτρα λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς χειριζόμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις ε, υποθέσεις προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια ανθρώπινη επανεισδοχή. Δεύτερον, σε ποιον βαθμό τα κράτη με τα οποία ε, πραγματοποιούμε επανεισδοχές είναι πρόθυμα να συνεργαστούν με μας, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ε, ακολουθήσουν μια συγκροτημένη οδό και τρίτον δεν θα ήταν απαραίτητο ορισμένα προγράμματα ένταξης και, και επανένταξης να συνδέονται με την ανθρωπιστική βοήθεια ώστε οι άνθρωποι αυτοί που επαναπατρίζονται να δέχονται κάποια μορφή βοήθειας στα χωριά στα οποία επιστρέφουν. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Μια προειδοποίηση για λόγους οργανωτικούς. Όταν έρθει ο υπουργό στις 16.45 θα πρέπει να του δώσουμε το λόγο. Και μετά λαμβάνει η χώρα ψηφοφορία και μετά θα αποχωρήσουν τα μέλη. Τι θα κάνω λοιπόν. Θα ακούσουμε πρώτα όλα τις ερωτήσεις για επανεισδοχή Ίσως να μην έχουμε χρόνο για πλήρες απαντήσεις. Θα υποβληθούν γραπτός ή θα ξανάρθει ο κύριος Ρίτε σε συγκεκριμένη συνεδρίαση για να απαντήσει. Βέβαια, ξέρω δεν είναι καθόλου ικανοποιητική κατάσταση, αλλά τι να κάνω. Ε, λόγω χρόνου. Περίπου ένα λεπτό σας παρακαλώ καθένας και ζητώ συγγνώμη που σας τριμώχνω έτσι. Κυρία Γκυγιώμη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση για τη συμφωνία με το Αφγανιστάν, για τη διαθέτηση που έγινε. Δεν ξέρω αν είναι ώρα κατάλληλη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα να πω ότι αυτή η διαθέτηση που έγινε ε, σκοπό έχει τη διευκόλυνση της επιστροφής των 80.000 Αφγανών περίπου που είναι σε κατάσταση παράτυπη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η ρύθμιση ε, υιοθετήθηκε στις 4 Οκτωβρίου την παραμονή δηλαδή της διάσκεψης των δωρητών για το Αφγανιστάν. Είναι δύσκολο να μην ε, κάνουμε τον παραλληλισμό για αυτή την τυχαία, άρα και σύμπτωση αυτών των δύο γεγονότων. Και δυστυχώς ε, έχει παραγωνιστεί πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη σύναψη αυτών των συμφωνιών, κάτι που μας ε, δυσαρεστεί όπως φαντάζεστε. Πώς φαντάζεστε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και πώς μπορούμε και εμείς να βρεθούμε στο επίκεντρο αυτών των τόσο σημαντικών αποφάσεων. Ευχαριστώ. Ιδού ένα παράδειγμα το πόσο σημαντικό είναι εδώ ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και λυπάμαι που σα τριμώχνω έτσι το χρόνο. Η κυρία Βέξτρομ, σα ευχαριστώ και σα ευχαριστούμε κύριε Ρούτε που ήρθατε το απόγευμα για να μα ενημερώσετε. Αναφερθήκατε φυσικά στη Συμφωνία Επανεισδοχή, αυτό είναι και το θέμα τη συζήτηση, αλλά αναφερθήκατε και σε άλλα θέματα, τη διακήρυξη και τη συμφωνία με την Τουρκία, για παράδειγμα. Και συμφωνώ που είπατε και χαίρομαι που ε, είπατε ότι θα πρέπει πρώτα να πληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις προκειμένου να λάβει η χώρα απελευθέρωση των θεωρήσεων. Τώρα το κλείσιμο ε, τις και πόσο θετικά αποτελέσματα είχε. Μόνο 43 ε, θανάτους φέτος σε σχέση με τον πολύ ψηλότερο αριθμό των θανάτων πέρυσι. Δεν είναι κοινικό να μιλάμε για κάτι τέτοιο όταν γνωρίζουμε ότι έχουμε φτάσει στο απόγειο φέτος ε, και ακόμη δεν έχει κλείσει η χρονιά, αλλά παρόλα αυτά έχουμε πάνω από 6.000 θανάτους ε, ε, στη Μεσόγειο. Η διαφορά είναι ότι κλείσαμε το, τη δίωδο από το Αιγαίο Πέλαγος, αλλά τώρα οι άνθρωποι θαλασσοπνίγονται ακολουθώντας τη, τη διέξοδο από την Τινησία, τη Λιβύη, γενικώ στη Βόρεια Αφρική η Μεσόγειος έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο υγρό τάφο. όχι απλώς υπάρχει κίνδυνος να γίνει. Είναι ήδη πια ένα υγρό νεκροταφείο η Μεσόγειος. Και για την Τουρκία. Το αναφέρατε, αλλά θα ήθελα λεπτομέρειες. Πόσους ε, πρόσφυγες ε, ε, τουρκικής προέλευσης ε, προβλέπετε να ζητήσουν άσυλο στην Ευρώπη, γιατί ένα Σουηδικό θα ήταν και τις προάλλες επισήμανε το κίνδυνο ε, να έχουμε μαζικές ε, εξόδους από την Τουρκία πολιτικών, ε, ακτιβιστών, δημοσιογράφων, ανθρώπων που θα ζητήσουν άσυλο ή ακτιβιστών από την ομάδα ΛΟΑΔ. Πώς βλέπετε αυτή την προοπτική και την κατάσταση. Κυρία Βιόρκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ομολογήσω ότι πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω την προσέγγιση σας. Και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασύλου εξαρτάται από τον αριθμό των ανθρώπων που επαναπατρίζουμε. Νομίζω ότι η νομιμοποίησή μας θίγεται από κάτι τέτοιο και δεν ενισχύεται από τους αριθμούς των ανθρώπων που επιστρέφουμε. Νομίζω ότι επικεντρώνεται την ενέργειά σας σε λάθος πράγματα. Έχουμε πάρει στραβό δρόμο. Θα πρέπει να επενδύσουμε σε καλύτερη υποδοχή των προσφύγων, όχι στην ε, επιστροφή τους. Και συμφωνώ με προλαλήσαντες ότι θα έχουμε όλο και περισσότερους ετούντες άσυλο από την Τουρκία. Ήδη έχουμε αύξητο αριθμό των προσφύγων από την Τουρκία, αλλά θα συνεχιστούν ε, οι εισρωέ από τη χώρα αυτή. Έχουμε συμφωνία επανειστοχή με την Τουρκία. Ε, σκοπεύουμε να στείλουμε πίσω αυτούς τους ανθρώπους που θα ζητήσουν άσυλο από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Αφγανιστάν αρνήθηκε μια συμφωνία επανεισδοχής με την Σουηδία και επικροτώ αυτή την απόφαση. Τι θα συμβεί όμως με τους ανθρώπους που την χάνουν κακομεταχείρισης, γιατί Άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ε, στην προσπάθεια αναγκαστικής επιστροφής. Τι γίνεται με όλους αυτούς. Ή τι γίνεται με την αδήλωτη εργασία. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, που, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που εργάζονται αδήλωτα στην Ευρώπη. Τι θα γίνει με αυτούς όταν συνεχιστούν οι επιστροφές. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον ε, κύριο Ήθελα να κάνω ολόκληρο λογίδριο, αλλά δυστυχώ μα πιέζει ο χρόνο. Οπότε θα πω ότι απλώ η ομάδα μου, η ΣΥΑΡΑ, συμφωνεί με το σχέδιο κοινή πορεία Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και Αφγανιστάν και τι όλε τι προσπάθειε σύναψη συμφωνιών επανεισδοχή με τρίτε χώρε. Έχω μία συγκεκριμένη ερώτηση. Πώ έχει η κατάσταση με τη Σομαλία. Θα γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι η Σομαλή είναι από τι μεγαλύτερε, ίσω η μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων που ζητούν ανθρωπιστική ε, βοήθεια και είναι οι ε, πρόσφυγες για ανθρωπιστικούς λόγους. Ε, πώς σκοπεύετε να δρομολογήσετε τη συμφωνία με τη Σομαλή, την επαναπατρισμό των Σομαλών στην πατρίδα τους. κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή, κύριε Ρίτε. Μας είπατε ότι έχετε καρδιά δεν το αμφισβητώ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πώς το θέμα των δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι κάτι που γίνεται σεβαστό. Πρόσφατα έχουμε αυτές οι συμφωνίες επανιστοχής που έχουν μέρημνα τον αριθμό πικών μιας χώρας που βρίσκονται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ενώσεω, ανεξάρτητα από το κράτος δικαίου που ισχύει στη χώρα τους από την οποία έρχονται. Μας είπατε ότι. μας διαβεβαιώνεται ότι όλοι αυτοί που επεστράφησαν είχαν εξαντλήσει δυνατότητε προσφυγή. Πώ το κάνατε αυτό, πώ φροντίζετε, πώ το καταφέρνετε. Ξέρουμε όλοι ότι οι διαδικασίε στα κράτη-μέλη είναι διαφορετικέ από χώρα σε χώρα. Γνωρίζουμε ότι το δικαίωμα ασύλου είναι σε, σε διαφορετικού ρυθμού σε κάθε χώρα. Ένα υπήκο επιστρέφει στην πατρίδα του συναρτήσει τι αναλύσει ενό κράτου μέλου. Αυτό σημαίνει ότι δεν γίνονται μέχρι, τελ, μέχρι τέλους σεβαστά τα δικαιώματά του. Ένα παράδειγμα, είμαι Γαλλίδα, θα υποδεχθούμε τον Υπουργό Εσωτερικών σύντομα. Εδώ και κάποιες μέρες ένας Σουδανός υπήκος απελάθη από το Σουδάν, από τη Γαλλία προς το Σουδάν. Ενώ δεν είχε εξαντλήσει τα δικαιώματά του όσον αφορά τη διαδικασία χορηγήσεως ασύλου και πολλαπλασιάζονται αυτά τα παραδείγματα. Θα ήθελα λοιπόν το θέμα των δικαιωμάτων να ξαναγίνει ένα θέμα στο επίκεντρο των συζητήσεων σας άκουσα, δεν άκουσα να λέτε κάτι τέτοιο, ακόμα και αν έχετε καρδιά. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαρτζεντίνη έχει το λόγο. Πριν θέσω το ερώτημά μου, θα ήθελα να καταλάβω κάτι, Πρόεδρε. Είχαμε δύο θέματα. Το ένα ήταν η εφαρμογή των συμφωνιών επανειστοχή σημείο 6, η κοινή προσέγγιση, η μελλοντική προσέγγιση που ακολουθούν είναι ξεχωριστά, διότι ακούω κάποιου να αναφέρουν το θέμα σαν θέμα του Αφγανιστάν. Δυστυχώ, λέει ο Πρόεδρο, πρέπει να ακούσουμε και τα δύο. Τότε μου λείπει η παρουσίαση του Γενικού Διευθυντού όσον αφορά την κοινή μελλοντική προσέγγιση. Και εμείς σαν συντονιστέ, ζητήσαμε αυτό να είναι διαφορετικό θέμα. Εγώ θα το καθυστερούσα, τα ανέβαλα αυτό, αντί να τα θέσουμε όλα με τη μία. Δεν είναι και δίκαιο, διότι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν είναι συμφωνία επανεισδοχή. Καλό λέει ο Πρόεδρο, αυτό ήθελα να καλύψω. Λοιπόν, να απαντήσω. Να πω επίσημα, δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο. Τι θα κάνω λοιπόν να δούμε και αν σας αρέσει αυτό που προτείνω. Έχουμε μέχρι 16 και 45 περιθώριο. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το όριο. Διότι θα πρέπει να ακούσουμε τον Υπουργό. Δεν μπορούμε για διάφορους οργανωτικούς λόγους δεν μπορούμε να το καθυστερήσουμε. Μετά έχουμε ψηφοφορία, δεν μπορεί να καθυστερήσει αυτή. Και μετά θα αποχωρήσουν οι παριστάμενοι. Θα ήταν άδικο για σας και τον κύριο Ρόιτε να βιαστούμε. Εγώ λέω να ακούσουμε τώρα όλες τις ερωτήσεις και όσον αφορά το ζήτημα του Αφγανιστάν, όπω είπε και η κυρία Γκυγιόμ, υπάρχει και άλλο θέμα που θέθετα. Πρέπει να ρωτήσουμε την νομική υπηρεσία ποια είναι η φύση τη συμφωνία και ποιο είναι ο ρόλο μα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το κατανοώ. Χρειαζόμαστε χρόνο αυτό να το αναλύσουμε. Λοιπόν, προτείνω όλοι να πάρετε 1,5 λεπτό στη διάθεσή σα να το έχετε, να υποβάλλετε τι ερωτήσει. Τώρα το συζήτησα με τη γραμματεία. Θα ξανακαλέσουμε μετά τον κύριο Ρίτε ζητώντας του συγγνώμη για αυτό που γίνεται για μια άλλη συνάντηση και θα πάρουμε και γραπτός πριν ξανάρθει κάποιες απαντήσεις για να έχουμε κάποιο βάρος και κάποια θεμέλια για τη συζήτηση και θα τα ξαναπούμε μαζί του. Αυτό προτείνω. Λοιπόν, θα επιστρέψουν στο θέμα του Αφγανιστάν συγκεκριμένα, λέει η κυρία Σαρτζεντίνη. Καλώ. Και θα γίνει και άλλη παρουσίαση, λέει ο πρόεδρο του κ. Ρίτε. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να ακουστούν όλε οι ερωτήσει και έτσι τουλάχιστον θα χρησιμοποιήσουμε σωστά το 45 λεπτό. Θα διατρέξω λοιπόν τον κατάλογο. Έχουμε 4-5 συναδέλφου ακόμα. 1,5 λεπτό ο καθένα. Ξεκινάμε από εσά και θα κλείσουμε την κυρία Σπινέλη μέχρι τις 16.45. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Σαρτζεντίνη. Για το Αφγανιστάν, να πω ένα πράγμα. Το εξή. Το Ευρωκοινοβούλιο στη συνθήκη έχει το δικαίωμα να αναφέρεται και να έχει λόγο όσον αφορά τις συμφωνίες επανεισδοχής. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θεωρούν ότι αυτή δεν είναι επίσημη συμφωνία επανεισδοχή, άρα δεν πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα, αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε ξεχωριστή συζήτηση σε αυτή την Επιτροπή. Αυτό διεξήχθη. Θα σταματήσω εδώ για την ώρα. Η μόνη συντομή μοναδική ερώτησή μου για την άλλη συμφωνία επανεισδοχή είναι η άλλη. Ο κύριο Ρίτε αναφέρθηκε συμφωνία με την Τουρκία. Νωρίτερα το απόγευμα είχαμε μια συνάντηση ATP, νημίσαμε για τα hot spots, όπου ένα συναδέλφο τη γενική Διευθύνσεω Home μα είπε ότι η Τουρκία έχει ακριβέστατο τρόπο ερμηνεία τη συμφωνία αυτή με την Τουρκία. Δηλαδή, εκείνοι οι οποίοι δεν είναι πλέον στα ελληνικά νησιά δεν μπορούν να επιστραφούν στην Τουρκία στην ανταλλαγή ένα προ ένα. Έτσι ερμηνεύετε και εσεί τη συμφωνία. Αυτό έχει κάπου γραφεί, το έχουμε διγραπτό κάπου. Διότι εγώ που τα παρακολουθώ εκ του σύνεγγυ αυτά τη συμφωνία με την Τουρκία, αυτό είναι καινοφανή πληροφορία και μου εξηγεί γιατί διστάζει τόσο κόσμο να μετακινήσει τους πρόσφυγες από τα νησιά προς την υπηρετική χώρα. Ευχαριστώ. Θα κάνω μια πρόταση στο τέλο. έτσι το επαναλαμβάνω. Η κυρία Άλμπιου έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι κατά τη γνώμη μου είναι επικίνδυνη αυτή η εισαγωγή που μας έκανε ο Γενικός Διευθυντής ε, εξηγώντα μας τη διαφορά μεταξύ των προσφύγων και των μεταναστών. Εμείς θεωρούμε ότι ο πρόσφυγας είναι εκείνος ε, που ε, καλύπτεται από την, από την Συμφωνία της Γενέβης και δικαιούται διεθνή προστασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο μετανάστης πρέπει να απελαθεί γιατί οι μετανάστες αυτοί που εσείς αποκαλείτε οικονομική μετανάστες, λες και ήταν ε, εθελοντική αυτή η προσπάθεια τους. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να γλιτώσουν από την πείνα, από τη φτώχεια. Δεν διαλέγουν τη μετανάστευση με την ελεύθερη τους βούληση. Είπατε επίση ότι θέλετε έτσι να σταματήσετε το δουλεμπόριο και το, τη σωματεμπορία. Αλλά και αυτό πόρο απέχει από την πραγματικότητα. Αν θέλετε να σταματήσετε τη λαροθροδιακίνηση και τη σωματεμπορία, θα έπρεπε να του εξασφαλίσετε τον τρόπο να διαμένουν και να εργάζονται νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο έτσι θα εξαρθρώνετε τα κυκλώματα τη λαροθροδιακίνηση και τη σωματεμπορία. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία με την Τουρκία, που φαίνεται ότι σα ικανοποιεί. Όντω, μειώθηκαν οι θάνατοι στο Αιγαίο, αλλά είχαμε ρεκόρ θανάτων στη Μεσόγειο, στην κεντρική Μεσόγειο και κυρίως ε, στις, ε, στο διάπλο από τη Λιβύη. Γιατί αυτό που καταφέρατε με την συμφωνία με την Τουρκία είναι να εξωθήσετε τους ε, πρόσφυγες σε πολύ πιο επικίνδυνες διόδους, κάτι που τους θαλασσοπνίγει στη Μεσόγειο. Ενώ αυτό που έπρεπε να κάνουμε για να αποφύγουμε τους θανάτους είναι να εξασφαλίσουμε νόμους διάβλους φαίνεται ότι δεν θέλετε αυτές ε, τις ε, αλλαγές. Θα προσπαθείτε να αποτρέψετε τους μετανάστες από το να έρχονται. Επίσης, τι γίνεται με τις χώρες που έχουν εμπόλεμη κατάσταση, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν. Επιστρέφετε τους ανθρώπους στις βόμβες. Στο Αφγανιστάν ε, έχουμε βία, εμπόλεμη κατάσταση. Έχουμε πάνω από χίλιους νεκρούς, 70 τρομοκρατικές επιθέσεις. Θεωρείτε το Αφγανιστάν ασφαλή χώρα στην οποία θεωρείτε σκόπιμο να επαναπατρίσετε κόσμο. Ευχαριστώ κυρία Αναγκόμης κύριε Ρούιτε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους και τον πρόεδρο που είπαν ότι έχει παρακαμφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς το ρόλο που θα έπρεπε να διαδραματίσει σε, αυτή, σε αυτές τις συμφωνίες δοχής. Είπατε ότι η συμφωνία Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αποφέρει αποτελέσματα διότι έπληξε τους, τους σωματεμπόρους. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ ήμουν 15 μέρες στην, ε, στην Ελλάδα και στα ε, σύνορα με την ε, Φύρομ και εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ε, διακινητές ανθρώπων και μάλιστα βγάζουν και περισσότερα κέρδη γιατί τα πράγματα έχουν γίνει πιο επικίνδυνα. Επίσης, συ, συγκρίνατε ε, τους ανθρώπους που πέθαναν στο Αιγαίο ε, πέρσι και φέτος. Μα ξεχάσατε διάφορους ε, παράγοντες που έχουν πάψει να υπάρχουν. Υπάρχουν 400.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν πνιγεί στην Μεσόγειο ακριβώς επειδή έκλεισε ο διάδρομος μέσω του Αιγαίου. Μπορεί να μας εξηγήσει η Κομισιόν Πώ, μια χώρα όπω η δική μου, η Πορτογαλία, που είναι τόσο ανοιχτή στο να υποδεχθεί γεζίδι ε, πρόσφυγες από αυτήν την κοινότητα. Πηγαίνουμε στην Ελλάδα και βλέπουμε να ζουν εκεί άνθρωποι στις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Και υπάρχουν ήδη καταχωρισμένοι άνθρωποι, 1600, και δεν έχει σταλεί ούτε ένα άνθρωπο στην Πορτογαλία. Ποια, πού είναι η προστασία των ανθρώπων. Πού είναι η προστασία των ανθρώπων όταν ε, γνωρίζουμε ότι ε, μιλούμε για πάνω από 10.000 ανήλικους ασυνόδευτους που ειναι η προστασια των ανθρωπων οταν γνωριζουμε εξαφανιστεί. Που μήπως τελικά τα ίδια τα κράτη-μέλη μετατρέπουν αυτούς τους ανθρώπους σε τρομοκράτες. Γιατί αυτό κάνουμε όταν τους αγνοούμε και τους αφήνουμε να ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Τους αφήνουμε στα χέρια των εγκληματιών και των τρομοκρατών. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Βίτμπεργκ. Tack herr ordförande. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, στα πλαίσια των συμφωνιών να δούμε τι είδους ανθρώπους ε, επιστρέφουμε. Γιατί μερικοί του άσυλο που τους έχουν ε, απορριφθεί οι αιτήσει και δύο φορές δεν έχουν πια, δεν υποφέρονται από το καθεστώς ασύλου. Γι' αυτό έχουμε τέτοιες συμφωνίες επαναπατρισμού, επανεισδοχής. Και σε ό,τι αφορά την Τουρκία, η Τουρκία έχει στείλει πολύ περισσότερους από όσους έχει δεχθεί πίσω. Και είπαμε να παγώσουμε τη συμφωνία. Αλλά τι θα γίνει τότε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοια συμφωνία επανεισδοχής. Και υπάρχει και το θέμα του Αφγανιστάν. Υπογράψαμε μια συμφωνία επανεισδοχής με το Αφγανιστάν. Και η Σουηδία έχει δεχτεί πάνω από 40.000 πρόσφυγες από το Αφγανιστάν σε άσυλο ε, και τώρα το Αφγανιστάν αρνείται την ε, επανεισδοχή. Τι γίνεται, υπάρχει συμφωνία ενισχύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφγανιστάν, γιατί κάπως παράδοξο ακούγεται όλο αυτό. Κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να παριθμίσω κάποια σημεία, κάποιες ανησυχίες που έχω. Πρώτα απ' όλα, συμφωνίες για αναπτυξιακή βοήθεια υπό των όρων της ρυθμίσεως των μεταναστευτικών ροών. Αυτή η διασύνδεση είναι ο λόγος για τον οποίο δεν είναι ξεκάθαρο, κύριε τι εννοείτε όταν μιλάτε για καλή συνεργασία ή όταν μιλάτε για ικανοποιητικά αποτελέσματα. Δεύτερο σημείο, ο παραγωνισμός ε, του Ευρωκοινοβουλίου από τις διαπραγματεύσεις και από τη σύναψη των συμφωνιών. Δεν είναι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο παραγωνίζεται, διότι γίνονται μέσω δηλώσεων αυτή της συμφωνία, αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια. Η συμφωνία μεταξύ Ιταλίας και Σουδάν ήταν μια συμφωνία απόλυτα μυστική. Το Ιταλικό Κοινοβούλιο δεν είχε κανένα λόγο άλλο που με ανησυχεί και θα ήθελα απάντηση. Το non-paper του Μαρτίου. Σχεδόν τελείωσα, πρόεδρε, τελείωσα. Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί εντοπίζονται ασφαλείς περιοχές στο Αφγανιστάν. Αναφέρεται σταθεροποίηση του Αφγανιστάν. Εγώ δεν πιστεύω ότι υφίσταται στο Αφγανιστάν αυτή η σταθεροποίηση. Δεν πιστεύω ότι είναι ασφαλής χώρα. Ποτέ πριν, όσο σήμερα, το Ισλαμικό κράτος και οι Ταλιμπάν δεν είχαν ε, ελέγξει τόσο μεγάλες, τόσα πολλά εδάφη στο Αφγανιστάν. Περισσότερα τώρα από, από το 2001. Μετά τους ε, Σύριους, ε, μετά τη Συρία, από το Αφγανιστάν μας έρχονται οι περισσότεροι πρόσφυγες διότι είναι μια χώρα που δεν είναι ασφαλής το Αφγανιστάν. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη από όλους τους συναδέλφους που έπρεπε να τους στριμώξω και να στριμώξω με τόσο σοβαρά θέματα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Έχω κάποιες προτάσεις. Απαντώ και σε αυτό και στον κύριο Ριούτε. Επομίζομαι τις ευθύνες. Δώσαμε μόνο μία ώρα σαν το θέμα. Θα έπρεπε να αρκεί, αλλά δεν αρκεί. Γιατί είναι πάρα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Διμερέ κιόλα, με δύο κομμάτια, δύο τμήματα. Πρόταση. Το κοινό μέλλον για το Αφγανιστάν, την κοινή προσέγγιση, θα το θέσουμε αυτό σαν ξεχωριστό θέμα όταν ξανάρθει ο κύριο Ρίτε. Θα τον προσκαλέσουμε το ταχύτερο δυνατόν. Φαίνεται ότι συμφωνεί, θα το συζητήσω μαζί του, θα το κανονίσω μετά τη συνεδρίαση, για να επιστρέψει και ο Ρίτε να το συζητήσουμε αυτό το δεύτερο τμήμα. Και μετά τι απαντήσει, τι ερωτήσει και τι συζητήσει στο πρώτο τμήμα. Εν τω μεταξύ, ίσω θα πρέπει να δοθούν και γραπτώ κάποιε απαντήσει. Είχαμε και προηγούμενο. Χρειάζονται περισσότερο χρόνο για απαντήσει ή ερωτήσει που έθεσαν οι 12 συνάδελφοι. Για το ερώτημα τη κυρία Γκυλιόν, το θέμα που έθεσε. Και το έθεσε η κυρία Σατζαντίνη και η Άννα Γκόμες και άλλοι. Δηλαδή συμφωνία με το Αφγανιστάν. Να ζητήσουμε την νομική υπηρεσία να το εξετάσει το θέμα και να αποφανθεί για να είμαστε σίγουροι ότι γίνονται σεβαστά τα προνόμια μας. Δεν είχαμε επίσημο ρόλο. Πρέπει λοιπόν αυτό να διλευκανθεί. Συμφωνεί να επανέλθει και ο Ζλούιτε να συζητεί το δεύτερο κομμάτι. Αν συμφωνείτε συνάδελφοι, αυτό θα κάνουμε. Το δεύτερο τμήμα της συζητήσεως για το Αφγανιστάν θα το συζητήσουμε ξανά με τον κύριο Ρίτε ταχύτερο δυνατόν. Έρχεται ο κύριος Υπουργό και γι' αυτό θέλω να ζητήσω. Ήρθε ο Υπουργό. Λοιπόν, να κάνει ένα-δύο σχόλια κύριε Ζουρίτε. Ακούσατε την πρότασή μου συνάδελφε. Συμφωνείτε, την ακούσατε. Συμφωνείτε. Δεν συμφωνείτε με, με δισταγμό έτσι, τέλος πάντων διστακτικά έτσι, με τα βία συμφωνείτε. τώρα θα πιστέψω και Ζουρίτε. Θέλετε τώρα να δώσετε κάποιες απαντήσεις για τα πιο σημαντικά θέματα, και Ζουρίτε. Γενικά σχόλια και μετά με τα χαράς να επανέλθω σε άλλη περίσταση και να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όλοι συμφωνούμε, χρειαζόμαστε μια σφαιρική, μια ληστική ε, προσέγγιση για τη μετανάστευση. Σήμερα Αναφέρθηκα στην επανεισδοχή, γιατί ήταν ένας από τους ε, πυλώνες και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να κατηγορήσει εμένα ή την Κομισιόν ότι δεν εξετάζουμε και τους άλλους ε, πυλώνες. Απλά δεν έχει νόημα να συζητούμε πάντοτε τα πάντα ε, μαζί. Δεύτερον, όσον αφορά ε, την ε, κατηγορία προς εμένα ότι αγνοούμε την κατάσταση ε, στην κεντρική μεσογειακή οδό. Πρέπει να σας πω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό που συμβαίνει εκεί είναι πραγματικά τρομακτικό, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να σας πω ότι οι ροές που έρχονται από την κεντρική Μεσόγειο όσον αφορά την εθνικότητα και την υπηκότητα είναι τελείως διαφορετικές από τις ροές εθνικοτήτων που έρχονται μέσω του Αιγαίου Πελάγους. Δεν ε, συνέκρινα καθόλου μάλιστα τις ε, δύο αυτές ε, περιπτώσεις. Για διάφορα άλλα θέματα πιστεύω ότι θα, πρέπει, θα χρειαστεί να γίνει μια λεπτομερέστερη συζήτηση. Μπορούμε να συζητήσουμε για την Κίνα, τη Σομαλία, μπορούμε να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες αν θέλετε. Θα ήθελα ε, να τα αφήσουμε εδώ, αλλά ε, ευχαρίστως να ξαναέρθω και να συζητήσουμε για τα ζητήματα της επανεισδοχής και συγκεκριμένα για το Αφγανιστάν, αλλά και ε, εν γέννη. Ωραία. Θα ξαναθέσουμε λοιπόν το θέμα του Αφγανιστάν σε ημερήσια διάταξη το συντομότερο δυνατό, για να έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε. Ένα μικρό διαλυματάκι θα κάνουμε και περνάμε αμέσως στο επόμενο θέμα μας.

Thank you, colleagues, Ευχαριστώ συνάδελφοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε το σημείο 7. Ανταλλαγή απόψε με τον Μπερνάρ Καζνεύ, Γάλλο Υπουργό Εσωτερικών. Χαίρομαι πολύ που βρίσκεται εδώ ε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Όπως γνωρίζετε, ο κύριος Καζνεύ έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Επιτροπή μας, καθώς στις διαπραγματεύσεις για το PNR είχε, με, είχε επιμέρους συναντήσεις με μέλη της Επιτροπής μας και πολύ συχνά συνεργάστηκε και με τους συντονιστές σε πολύ δύσκολες συζητήσεις και το λέω γιατί είναι ένας από τους υπουργούς που πολύ συχνά έχει συνεργασία και επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για προφανώς αμφιλεγόμενα ζητήματα, φλέγοντα ζητήματα αλλά είναι γεγονός ότι τουλάχιστον μας αφιερώνει τον χρόνο του και το εκτιμούμε πολύ αυτό. Σήμερα λοιπόν θα συζητήσουμε για πολλά από αυτά τα θέματα, για το πού βρισκόμαστε. Έχουμε και ένα πλαίσιο, έχουμε μια ε, ψηφοφορία σήμερα για την οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, έχουμε τον κώδικα συνόρων Σέγγερ, ε, ένα, ε, ένα ε, θέμα για τον μηχανισμό αναστολής θεωρήσεων. Πολύ συχνά έχουμε συζητήσει εδώ την κατάσταση στο Καλέ σε συνεδριάσεις τη Επιτροπής μας. Είναι μια σειρά από ζητήματα καθόλου εύκολα με τα οποία ασχολείστε εσείς, αλλά τα συζητούμε όπως είπα και εμείς εδώ στην Επιτροπή μας και θεωρήσαμε ότι ήταν κατάλληλη στιγμή για να γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψε με εσάς. Στο πλαίσιο αυτό των σχέσεων και όλας που έχετε αναπτύξει με επιμέρους μέλη της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για αυτό και για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Θα ε, ξεκινήσουμε. Ε, σας δίνω 15 λεπτά κύριε Υπουργέ. Στη συνέχεια θα πάρουμε ερωτήσεις και τοποθετήσει. Σας καλωσορίζω λοιπόν. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ και έχετε τον λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι Αντιπρόεδροι και μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω θερμότατα για την υποδοχή και τη φιλοξενία σας εδώ στην Επιτροπή. Μάλιστα, είχα την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να έρθω αρκετές φορές στην Επιτροπή σας, ιδιαίτερα μετά τα τραγικά συμβάντα που βήθησα στο πένθο στη Γαλλική Πρωτεύουσα το 2015 και μάλιστα και τότε με υποδεχθήκατε θερμά για να εγγύψουμε σε μία σειρά θεμάτων που ε, εδώ και καιρό σας απασχολούσαν το θέμα του Μητρώου των Στοιχείων Επιβατών, του PNR, το θέμα του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία και πάλι να σχολιάσω αυτά τα θέματα στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι μόνο τη Επιτροπή σα, αλλά και των άλλων Επιτροπών, για την ελεγγύη που έδειξαν προ τη χώρα μου, προ την πατρίδα μου, όταν επλήγει δρυμύτατα από τι τρομοκρατικέ επιθέσει. Ε, και σήμερα και το 2015, αλλά και το καλοκαίρι του 2016. Για παράδειγμα, την τραγωδία τη Νίκαια, ε, τη δολοφονία ε, δύο αστυνομικών στη Μανιαβίλη και τη δολοφονία ενός ιερέως σε μια πόλη της Γαλλίας. Πάνω από 230 άτομα έχασαν τη ε, ζωή τους στη Γαλλία τα τελευταία, στους τελευταίους μήνες ε, και πολλές χιλιάδες έμειναν τραυματίες σε αυτόν τον ε, αποτρόπιων τρομοκρατικών επιθέσεων που χτύπησαν τη Γαλλία και το Βερίο και άλλες χώρες. Εκτιμώ ιδιαίτερα την υποστήριξή σας και Εκτιμήσαμε ιδιαίτερο στο γεγονός που, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ενέκυψε στα θέματα αυτά που ήταν αντικείμενο τριμερών διαλόγων και ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει κατεπηγόντως κάποια κέρια ζητήματα. Αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα και την τρομοκρατία αλλά και τη μεταναστευτική κρίση με σημαντικό αριθμό αφήξεων. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, περίπου ένα εκατομμύριο και τους τελευταίους 18 μήνες, πρόκειται για μετανάστες και πρόσφυγες που οι περισσότεροι προσπάθησαν να γλιτώσουν από εχθροπραξίες, βία, διώξεις στις πατρίδες τους. Μερικές φορές προσπάθησαν να γλιτώσουν από την αθλειότητα, τη φτώχεια και έχουν καταφτάσει στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Έχουμε τώρα δύο διαφορετικά θέματα, το θέμα της τρομοκρατίας και το θέμα της μετανάστευσης. Μερικοί κάνουν αυτό το αμάλγαμα μεταξύ των δύο, το, τα συγχαίων, τα συνδέουν για πολιτικούς λόγους. Εμείς ε, δεν συνδέουμε αυτά τα δύο θέματα, τα διαχωρίζουμε, αλλά πιστεύω θα πρέπει να επαγρυπνούμε ώστε ο έλεγχος στα εξωτερικά σύνορα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι αποτελεσματικός και να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ώστε να μπορούμε να υποδεχόμαστε όσους ε, θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί νιώθουν ότι διώκονται στις πατρίδες τους. Έχουμε λοιπόν δύο κατεπήγοντα θέματα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Και για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο καταπήγοντα θέματα δεν θα πρέπει να αρκόμαστε σε λογίδρια, διακηρύξεις ε, και αγαθές προθέσεις. Θα πρέπει να δράσουμε πάρα αυτά με αποφασιστικότητα και πυγμή για να αποδείξουμε και εμπράκτος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να δώσει αποτελεσματικές ε, λύσεις και απαντήσεις στις δύο προκλήσεις που προβληματίζουν τους συμπολίτε μας. Και γι' αυτό ακριβώ συμφωνήσαμε το οδικό χάρτη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μπρατισλάβα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος ε, για να καθησυχάσουμε και να πείσουμε τους συμπολίτε μας που έχουν πολλές αμφιβολίες ε, γιατί όλο και περισσότεροι συμπολίτε μας ε, αμφιβάλλουν για το κατά πόσο είμαστε αποτελεσματικοί και δεν μπορούμε παρά να προβληματιζόμαστε για αυτή την απόσταση και το χάσμα που δημιουργείται μεταξύ πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο για να ανακτήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μόνο υπό τον όρο ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ε, συντονίζονται και με ειλικρινή και διαφανή διάλογο μεταξύ Συμβουλίου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να συντονιστούμε. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Θα πρέπει να αναλάβουμε συγκεκριμένα μέτρα στα πλαίσια της συναπόφασης και με διαρκή διάλογο που μας τον επιβάλλουν οι συνθήκες. Και μάλιστα αυτός ο διάλογος είναι η καλύτερη μέθοδος για να καταλήξουμε σε ισορροπημένες πολιτικές. Και ως Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ε, θα ήθελα φυσικά να ενισχύσουμε αυτό το διαθεσμικό διάλογο και να έχουμε και άμεσες ε, ανταλλαγές απόψεων και πιο γενικές μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Αυτό κάνουμε σήμερα και αυτό είχαμε κάνει και το Φεβρουάριο του 2015 όταν είχα ξανάρθει. Και θα ήθελα να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί πραγματικά ε, είναι επιτακτική ανάγκη άμεση ανάληψη δράσης, γιατί καθημερινά διαπιστώνω πόσο σοβαρά είναι τα θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στα κοινοτικά θεσμικά όργανα και στην ικανότητά τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Μάλιστα είχαμε πολύ σημαντική πρόοδο από κοινού την ε, υλοποιήσαμε τους τελευταίους 18 μήνες και αυτή η πρόοδος ε, αποτελεί την απόδειξη της ικανότητας να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το κινητήριο ομοχλώ τον πρωταγωνιστικό του ρόλο και τι σημαντικέ πρωτοβουλίε που ανέλαβε και ευχαριστώ και την Επιτροπή σα για τα ε, εντυπωσιακά αποτελέσματα. Γι' αυτό ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε πρώτα πλήρω τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι απαραίτητο για να μα προστατεύσει από την τρομοκρατική απειλή και να διαχειριστούμε πιο αποτελεσματικά τι αυξανόμενε μεταναστευτικέ ροές, που δεν πρόκειται να μειωθούν του επόμενου μήνε. Ε, το αντίθετο, μάλιστα ε, παραμένουν αμύωτε οι μεταναστευτικέ ροέ, ακόμη και κατά τη χειμερινή περίοδο και από τη Μεσόγειο ακόμη, που σημαίνει ότι το φαινόμενο είναι διαρθρωτικό, έχει διαρθρωτικό χαρακτήρα. Θα πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε αυτό να το έχουμε κατά νου. Και αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τον πλήρη έλεγχο των εξωτερικών συνόρων με αποτελεσματικό και οργανωμένο τρόπο. Γι' αυτό και έληφθησα πολλά σημαντικά μέτρα χάρη αυτή τη διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων. Και χαίρομαι, τον περασμένο Απρίλιο καταλήξαμε σε συμφωνία ε, επί της οδηγίας ε, για ένα, για ένα μητρό των ε, στοιχείων επιβατών των αεροπορικών εταιριών, το λεγόμενο PNR. Μάλιστα, το, ήδη το Φεβρουάριο του 2015 είχαμε πολλές απορίες και πολλές υποψίες κατά του PNR και πολλοί ευρωβουλευτές θεωρούσαν ότι το ευρωπαϊκό PNR ε, διασφάλιζε κάποια ασφάλεια, αρκεί να ε, εφαρμοζόταν ε, ταυτόχρονα από όλε χώρε, αλλά δημιουργούσε κάποια προβλήματα προστασία προσωπικών δεδομένων. Αλλά καταλήξαμε σε μια καλή ισορροπία, υπό τον όρο όμω ότι θα δοθεί μια συνέχεια και ότι τα κράτη-μέλη θα εφαρμόσουν το PNR με βάση του στόχου που έχουν αναλάβει και τι υποσχέσει που έχουν δώσει και μάλιστα ήδη έχουμε το δικό μας σύστημα PNR και την αρμόδια μονάδα για τους ε, επιβάτες που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή της πρότασης του PNR και θα θέλαμε για τις ενδοκοινωτικές πτήσεις και τις ε, πτήσεις charter το PNR να λαμβάνει υπόψη τις διάφορες επιλογές γιατί αν δεν το κάνουμε θα χάσουμε την αποτελεσματικότητα αυτού του μηχανισμού. Ε, και τους ε, στόχους ε, της ασφάλειας. Δεύτερο θέμα, η, η ανανέωση της Frontex για την προστασία των συνόρων και στο συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Έχουμε πλέον 1.600 ε, υπαλλήλους που μπορούν να κινητοποιηθούν για τα εξωτερικά σύνορα και μάλιστα μέσα σε 6 μήνες σε χρόνο ρεκόρ υιοθετήσαμε τη νέα πρόταση και η Γαλλία συμβάλλει στη Frontex έχει ε, αποσπάσει 170 υπαλλήλου στη Frontex και θα εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα μέσα για να στεφτεί με επιτυχία η αποστολή τη Frontex. Και μάλιστα είχα παρελειμμένο την ευκαιρία να τονίσω την επιθυμία της Γαλλίας να οργανωθεί μια άσκηση σε πραγματικές ε, συνθήκες ε, μεγάλων διαστάσεων σε συνεργασία με τον, τον Υπουργό της Γερμανίας Νταμεζιέρ και Εκεί θα πρέπει να δούμε το προσωπικό που κινητοποιείται, τις συνεισφορές των ε, χωρών μελών και πόσες δυνάμεις κινητοποιούνται ώστε να εξασφαλιστεί επί τόπου αποτελεσματικός έλεγχος. Frontex, PNR και ένα τρίτο θέμα που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ο κώδικας των συνόρων Schengen για να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός έλεγχος των εξωτερικών συνόρων. Αυτό είναι προτεραιότητα εξαιτία του υψηλού επίπεδου απειλής που αντιμετωπίζουμε, ειδικά στη Γαλλία. Εδώ και ένα χρόνο ζητούσαμε την ε, επαναφορά των σύνορων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τι τρομοκρατικέ επιθέσει του 2015. Πρόκειται για ένα απαραίτητο μέτρο και στο ισχύον πλαίσιο που θα πρέπει να διατηρηθεί, να μείνει εν ενεργεία στο μέτρο που το απαιτούν οι συνθήκε και άλλα κράτη-μέλη χρειάστηκε να λάβουν παρόμοια μέτρα για να αντιμετωπίσουν τι έκτακτες μεταναστευτικέ ωραίε και χαιρετίζω την ικανότητα αντίδραση που έδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να επιτρέψει τα κρατη να αντιμετωπίσουν άνευ προηγουμένου καταστάσει. Ε, επαναφέροντας αυτούς τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα. Επίσης θα πρέπει ε, να εφαρμόσουμε και πάλι ε, την, το χώρο ελεύθερης διακίνησης σε ένα όμως πλαίσιο ασφάλειας και μετανάστες που εξελίσσεται ραγδαία. Και γι' αυτό ακριβώς ε, εκφράζω την επιθυμία μέχρι τα τέλη του έτους να καταλήξουμε στη συμφωνία για το νέο κείμενο και νομίζω ότι η Γαλλία έχει επιδείξει συνεργάσιμο και διαλλακτικό πνεύμα και ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει το ίδιο. Μάλιστα, ε, αυτά ήταν από τα σημαντικά θετικά βήματα που κάναμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη και κάποια, ε, το γεγονό ότι κάποια νέα στοιχεία είναι ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν την έκτακτη κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι και πιο άμεση την αντίδρασή μας. Η Γαλλία προσπάθησε να αντιμετωπίσει ε, και τα, τις προκλήσεις ασφάλειας και τις προκλήσεις μετανάστευσης και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια τους τελευταίους 18 μήνες ε, υιοθετήσαμε ε, δρακόντια μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πρωτόγνωρες απειλές. Αυξήσαμε τι δυνάμει ασφαλεία και εσωτερική τάξη και τι μυστικέ υπηρεσίε. Αυξήθηκε κατά 20% και ο προπολογισμό του. Υιοθετήσαμε και νέα νομοθετικά μέτρα, για παράδειγμα το νόμο για τις μυστικές υπηρεσίες. Μάλιστα κάποιοι βουλευτές ε, ε, έθεσαν απορίες για το κατά πόσο είναι συνταγματικός αυτός, αυτός ο νόμος. Επίσης, ε, έχουμε μια νέα επιτροπή υπατιαρχή που αποφαίνεται επί της ενεργοποίησης των νέων τεχνικών μυστικών υπηρεσιών. Έχουμε και το νόμο της 13η Νευρίου 2014 για να μπλοκαριστούν ε, διοικητικά κάποιες ιστοσελίδες του ίντερνετ ε, και μάλιστα συνεργαστήκαμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αποσύρουμε κάποιες ιστοσελίδες που προωθούσαν την δημοκρατία και έχουμε και το νόμο του 2016, Ιουνίου 2016 που επιβάλλει κάποια μέτρα ε, για την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να εξασφαλίσει με βάση το, το δίκαιο ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Ε, φυσικά υπάρχει και το, η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, δεν μπορούμε να το αποσιωπήσουμε αυτό. Ε, ξέρω ότι έχει δημιουργήσει προβληματισμούς και ερωτηματικά. Θεσπίστηκε αυτή η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να μπορέσουμε με κάποια μέτρα διοικητικές αστυνομίε και κάποιες, ε, ε, κάποιους ελέγχους κατοίκων και κρατήσεις κατοίκων να, αποφασ... να λάβουμε αυτά τα μέτρα από τη διοίκηση υπό τον αυστηρό έλεγχο ε, ενός ε, διοικητικού δικαστή και μάλιστα είχαμε μία από τις σημαντικότερες συνομολογίες ε, διοικητικών δικαστών που μιλούν για, την, για το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και μάλιστα είχαμε την απόφαση Μπεζαμά του 33 και του 1962 και πολλέ αποφάσει της διοικητική αστυνομία αφισβητήθηκαν από το διοικητικό δικαστή κατά την εφαρμογή των διατάξεων τη κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν κακέ οι αποφάσεις, ήταν ελάχιστε οι αποφάσει που αφισβητήθηκαν, αλλά σα διαβεβαιώ ότι υπάρχει δικαστικό έλεγχο αυτών των αποφάσεων τη αστυνομική δικαιοσύνη, και μάλιστα με πολύ αυστηρό τρόπο και μάλιστα με την κατάσταση εκτάκτου ανάγκη. μπόρεσαν οι, οι διοικητικέ να κάνουν κατάσχεση σημαντικού αριθμού όπλων και μάλιστα ε, ε, συλλάβαμε υπόπτους ε, που θα διέπραταν τρομοκρατικές ενέργειες και που είχαν στην κατοχή του όπλα. Έχουμε κινητοποιηθεί λοιπόν για το θέμα αυτό. Και να πω και δύο λόγια για τη μεταναστευτική κρίση. Την ανέφερα στα πλαίσια της, του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων που έχουμε θεσπίσει. Λοιπόν, Ήθελα να αναφερθώ σε κάποιε αποφάσει που λάβαμε στα πλαίσια του γαλλικού δικαίου και σε διάφορε τοποθεσίε τη Γαλλία όπου ετίθεται το πρόβλημα το μεταναστευτικό και κυρίω στο Καλέ, όπου υπήρχαν πάρα πολλά ερωτηματικά εκεί και προβλήματα. Έγινε σημαντική επιχείρηση. Θα ήθελα να πω κάποια λόγια στην Επιτροπή σα. Καταρχά, πήραμε αποφάσει να αφορά το άσυλο, την πολιτική ασύλου. Θεωρούμε ότι αν θέλουμε να μπορέσουμε εκείνου για εκείνου που δικαιούνται άσυλο, για να μπορούμε να προστατεύσουμε αυτούς που έχουν δικαίωμα ασύλου, πρέπει να μπορούμε να επαναπατρίσουμε αυτούς που δεν δικαιούνται ασύλου. Άρα θα πρέπει να έχουμε σωστή πολιτική ασύλου και αυτό θα μειώσει και την, ε, την εξέταση των αιτήσεων ασύλου, θέτοντας τη διάθεση των δικήσεων που είναι επιφορτισμένες με αυτή την επεξεργασία τα ανθρώπινα μέσα και τον προπολογισμό για το κάνουν. Αυτό εξαρτάται βέβαια και από τι δυνατότητε που έχουμε, δηλαδή να δημιουργήσουμε τι ε, δυνατότητε στέγαση για να επιτρέπουν να γίνεται αυτή η επεξεργασία του τίματο ανθρώπινε συνθήκε που αντιστοιχεί στην προσέγγιση που έχει η χώρα μα όσον αφορά ε, τι θεμελιώδει αρχέ. Από αυτή την άποψη έχουμε αυξήσει πάρα πολύ σημαντικά το αναγκαίο προσωπικό Μέσο όρο ετήσεως ασύλου ήταν 24 μήνε και είναι 18, πήγε σε 14 μήνες επεξεργασία αιτήματο άσυλου και θα μεθάσουν στου 9 μήνε. Επίση, βελτιώσαμε τα κέντρα υποδοχή των ετούντων άσυλο. Είχαμε 22.000 όταν είχε έρθει στην εξουσία. Τώρα έχουμε 42.000 ε, και έχουμε ολοκληρώσει τον όλο μηχανισμό μέσω πολιτικών στέγασης κατεπίγουσες ε, φροντίδες για στέγαση για να στεγάζονται τα άτομα που είναι τούντε άσυλο και αντιμετωπίζουν δυσκολίε. Λοιπόν, βελτιώνουμε τα μέσα, μειώνουμε τη διάρκεια επεξεργασία των ετοιμάτων ασύλου και θέλουμε η απομάκρυνση των ανθρώπων να γίνεται με αξιοπρεπεί όρου, εκείνων που δεν την χάνουν δικαιώματο ασύλου. Συζητείτε και το άλλο, ότι ε, στέλνουμε πίσω λιγότερου ανθρώπου ε, από τα σύνορα από ό,τι πριν. Στα πλαίσια λοιπόν των μεθορικών ελέγχων μπορέσαμε να εφαρμόσουμε τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες στα σύνορα, περίπου 50.000 ανθρώπους στείλαμε το 2006 στην πατρίδα τους, στα σύνορα. Και αν το λάβουμε υπόψη αυτό, έχουμε ισορροπημένη πολιτική. Δεχόμαστε αυτούς που θα πρέπει να δεχτούμε και γίνεται επαναπατρισμό σε εκείνους που δεν μπορούμε να δεχτούμε, σεβόμενοι πάντα με αυστηρότητα τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να πω κάτι για το καλέ. Ε, στο καλέ εδώ και δεκαετίες... Λοιπόν, στη βόρεια ακτή, στο Καλέ και αλλού, στο Σενγκάτ, το παρελθόν είχαμε συγκέντρωση μεταναστευτών που ήταν στα χέρια των διακινητών και ήθελαν να πάνε στην Βρετανία, χωρίς να ζητάνε άσυλο στη Γαλλία. Ήταν σαφής η πολιτική μας. Αντί να αφήσουμε λοιπόν αυτούς τους μετανάστες που 80% αυτών ε, θα, έπρεπε να προστατευτούν ε, στη Γαλλία, ή στην Ευρώπη, αντί να τα αφήσουμε, αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους στα χέρια των διακινητών στο Καλέ, διαλύσαμε λοιπόν τα δίκτυα, κάθε χρόνο 20% περισσότερα δίκτυα διαλύαμε το 2014, διακινητών, δίκτυα διακινητών. Και έτσι στο Καλέ συγκεντρώσαμε τι δυνάμει ασφαλεία, διάφορε μονέ αστυνομία, για να διαλύσουμε αυτά τα μαφιόζικα δίκτυα που ασχολούνταν με το εμπόριο ανθρώπων. Μετά θελήσαμε και κάτι άλλο να πετύχουμε. Εκείνοι που ήθελαν να πάνε στη Βρετανία από τη στιγμή που δεν μπορούν να περάσουν για λόγους που αφορούν στη σύμβαση που είχαμε υπογράψει ε, η προκάτοχή μου, τη συμφωνία που είχε υπογραφεί, για αποτρο... να αποτραπεί η διέλευση των μεταναστών προς τη Βρετανία, εφαρμόσαμε τις συμφωνίες. Όταν υπογράφουμε συμφωνίες, ε, τις σεβόμαστε. Λοιπόν, θέλουμε να σεβαστούμε λοιπόν τις συμφωνίες και γι' αυτό κινηθήκαμε το τρόπους. Ως υπεύθυνη χώρα αποφασίσαμε λοιπόν αυτούς τους μετανάστευς να τους ε, διηγήσουμε στο να ζητήσουν άσυλο στη Γαλλία, αντί να τους αφήσουμε στα χέρια των διακινητών. Από τη στιγμή που αποφασίσαμε αυτή τη στρατηγική δεν θα έπρεπε να τους αφήσουμε στο καλέ, θα έπρεπε να πάνε σε κέντρα ε, υποδοχής πιο σωστά, να μην είναι ευάλωτοι, να πάνε σε σωστά κέντρα υποδοχής. Θέλαμε. Λοιπόν, 465 κέντρα υποδοχής υπάρχουν και στους 18 μήνες. Περίπου 13.000 άνθρωποι από το Καλέ πήγαν εκεί. 2.000 ε, ασυνόδευτα παιδιά μεταξύ αυτών που πήγαν σε ειδικά κέντρα για τους ανήλικες και εξετάζεται και η υπόθεση αυτών και από την ε, Βρετανία για να δουν κατά πόσο αυτά τα παιδιά μπορούν να γίνουν δεκτά στη Βρετανία στα πλαίσια της εφαρμογής των κανόνων του α, ε, Δουβλίνου. Λοιπόν, ανέλαβε η Γαλλία την υποδοχή 13.000 ανθρώπων στα κέντρα υποδοχής προσανατολισμού και, στη, και περίπου 11.000 εκτός από τα απομονωμένα παιδιά να μπουν στο μηχανισμό χορηγής ασύλου και θα πρέπει τώρα να απομιστεί τις ευθύνες της η Βρετανία. Διότι είναι άνθρωποι που ήθελαν να πάνε ζητήσουν άσυλο στην Βρετανία και τους είχαμε δεχτεί στην Γαλλία, σύμφωνα με τις αρχές μας. Αλλά τα απομονωμένα παιδιά, τα ανήλικα παιδιά, από τη στιγμή που έχουν σχέσεις με τη Βρετανία, θα πρέπει λοιπόν να τα υποφορτιστεί η ε, Βρετανία, σύμφωνα με την ομοθεσία τη Βρετανική. Λοιπόν, η Ιρλανδία, ενώ δεν ήταν υποχρεωμένη, σε ευχαριστώ γι' αυτό, υπέγραψε ένα νόμο που, σύμφωνα τον οποίο θα υποδεχτούν στην Ιρλανδία 200 ανήλικα παιδιά τους επόμενους μήνες. Να πω κάποια λόγια για να ολοκληρώσω να αναφερθώ σε αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Θέλουμε να λειτουργήσει ο μηχανισμός μετεγκατάστασης και είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσης που συνέβαλε σε αυτό. Περίπου τα δύο τρίτα των μετεγκατασταθέντων τους ε, δεχτήκαμε από τα hot spots. Θα θέλαμε αυτή η δουλειά να συνεχιστεί στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, στα στοιχεία η Γαλλία. Όσον αφορά τη δικασια μετεγκαταστασης μετεκατάστασης-εγκατάστασης, 4.240 κέντρα υποδοχής έχουμε. Έχουμε 2.500 περίπου ανθρώπους μου δεχτεί και πάνω από 35.000 αυτών που μετακαταστήθηκαν από την Ελλάδα ήρθαν στη Γαλλία. Οπότε η χώρα μας παίζει το ρόλο της όσον αφορά τη μετεκατάσταση και παίζει το ρόλο της και στο καλέ και θα συνεχίσει να το κάνει. Να πω κάποια θέματα όσον αφορά τις θεωρήσεις για την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Θα γίνει αυτό από τη στιγμή που θα υπάρξει ρήτρα διαφύλαξη. Αν δεν υπάρξει, δεν θα αναπτυχθεί ανεξέλεκτα αυτή η πολιτική, διότι αν γίνει κάτι τέτοιο υπονομεύουμε την ελεύθερη διακίνηση που είναι και το πνεύμα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσης, άρα πρέπει να εφαρμόζεται τη ρήτρα διαφύλαξης. Αυτό είναι ο όρος για την αποδοχή του προτινόμενου μηχανισμού για την απελευθέρωση από τις θεωρήσεις για τις χώρες που ζητούν κάτι τέτοιο Συμφωνούμε με το, με μηχανισμό αιτίας που ακολουθεί τη σωστή κατεύθυνση. Θα εξασφαλίζει και την σωστή ασφάλεια. Για το σύστημα εισόδου-εξόδου συμφωνούμε ε, και λαμβάνοντας υπόψη τον τρομοκρατικό κίνδυνο εάν δεν έχουμε τον κατάλληλο μηχανισμό για είσοδο-εξόδου και να, μπορούμε να διαπιστώνουμε τι γίνεται σε όλα τα σύνορα που τα οποία διέρχονται εκείνοι που ωφελούνται από τον μηχανισμό θα χάσουμε σημαντικά σε επίπεδο ασφαλείας και θα, εκτεθούμε, θα εκτεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κινδύνους οι οποίοι θα είναι πάρα πολύ σημαντικοί που θα υπονομεύσουν μακροπρόθεσμα την εφαρμογή των πολιτικών που είναι υποφελής για τους πολίτες, την ελεύθερη διακίνηση. Είμαστε λοιπόν, θέλουμε πάρα πολύ την οδηγία να εφαρμόσουμε κατά της και κάπου να καταλέξει η οδηγία κατά, για τον έλεγχο των όπλων. Λοιπόν, ανησυχούμε για την πορεία των συζητήσεων, για τα αυτόματα όπλα. Αυτό που προτείνεται είναι πάρα πολύ ευέλικτο, πολύ χαλαρό, πολύ φιλελεύθερο όσον αφορά τον κίνδυνο που εκπροσωπούν αυτά τα όπλα, κυρίως στα χέρια των τρομοκρατών. Οι εξαιρέσει οι οποίες προβλέπονται μπορούν και αυτές για χώρες όπου δικαιολογείται αυτό για λόγους ασφαλείας αποδοχή χρήση αυτών των όπλων από τους πολίτες για να υπερασπιστούν για την ασφάλειά τους, για να υπερασπιστούμε την ασφάλεια των πολιτών, αυτό δημιουργεί πρόβλημα διάδοσης των όπλων. Και μπορεί να πέσει στα χέρια τρομοκρατικών ομάδων και αυτό είναι πρόβλημα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο, διότι έχω πάρα πολλά πράγματα να πω και νομίζω ότι υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να μπορούμε να συνομιλήσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για την ευρύτατη παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Σχεδόν όλοι όσοι παρευρίσκονται στην αίθουσα έχουν ζητήσει το λόγο. Ε, ξανακοιτάω γιατί αλλιώς θα κλείσω τον κατάλογο ομιλητών. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις ε, κύριε Υπουργέ, ε, οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να μην μιλήσουν πάνω από ένα λεπτό ο καθένας ή δυνατόν, για να μπορέσουμε να λάβουμε και τις απαντήσεις από τον Υπουργό. Εντάξει, λίγο παραπάνω από ένα λεπτό, αν πραγματικά είναι απόλυτη ανάγκη, αλλά καταλαβαίνετε. Δεν είναι όλοι οι συντονιστές μα εδώ, οπότε θα λάβουν το λόγο οι συνάδελφοι με, τον, ε, με τη σειρά που τον ζήτησαν, την μέρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον Γάλλο Υπουργέ που επανειλημμένος ε, έχει έρθει στην Επιτροπή μας. Θα ήθελα πρώτα να σας εκφράσω την κατανόησή μου και την αλληλεγγύη μου. Την αλληλεγγύη μου για την ασφάλεια των Γάλλων και την ασφάλεια των Ευρωπαίων γενικώ. Σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο που μπλοκάρει η Γαλλία. Ένα ιδιαίτερο θέμα που μπλοκάρει η Γαλλία. Είμαι ο εισηγητή για τις θεωρήσεις και τους μηχανισμούς αναστολής και τους μηχανισμούς αμοιβαιότητας. Ε, ο κανονισμός 539 του 2001. Ε, μερικά θέματα είναι προφανή, αλλά καλό θα ήταν να τα τονίσουμε και πάλι. Όσο εγώ θα είμαι εισηγητής μιας έκθεσης, θα υποστηρίζω με νύχια και με δόντια το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη. Γιατί αυτό το ρόλο του συνομοθέτη προσπαθεί να αποδυναμώσει το Συμβούλιο. Εγώ πάντως θα τον προσπίσω αυτό το ρόλο με νύχια και με δόντια σε ό,τι αφορά το μηχανισμό αναστολής. Το πεδίο διαπραγμάτευσης είναι ο τριμερής διάλογος. Είναι γνωστό της πάσης. Οπότε ο εισηγητής, ο υποφερόμενος δηλαδή, θα διαπραγματευτεί ε, με την εκπεριτροπής προεδρία. Και φυσικά διαπραγματεύομαι και με τους συναδέλφους και ακούω τα πάντα, όλες τις γλώσσες, αλλά ο συνομιλητής μου θα είναι μόνο ο προεδρεύων Συμβουλίου. Δεν μπορούμε ε, να αντιμετωπίζουμε την α ή β φαϊνίδια της α ή β χώρας. Ε, γιατί τελικά καταλήγουμε σε μπλοκάρισμα όταν συνομιλητής μας δεν είναι μόνο ο εκάστοτε προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι άλλο θέμα. Ε, η κατάσταση στην οποία έχουμε προσκρούσει στο θέμα του μηχανισμού αναστολής. Έτσι, χώρες όπως η Γεωργία, η Ουκρανία, το Κωσυφοπαίδιο γιατί έχει δημιουργηθεί συνάρτηση με την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Και αυτή η εβδομάδα ελπίζω να είναι η τελευταία διορία για να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα έχω, συμφωνία, θα έχω συνάντηση με τους κοιόδης ηγητές την Τετάρτη, οπότε αν η Γαλλία αποφασίσει και δεήσει να άρει το βέτο της, Πιστεύω θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε την Πέμπτη το πρωί στην Επιτροπή, ώστε να μεταφερθεί αυτή η έκθεση στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Αν αυτό θα ήταν το θετικό σενάριο, αν δείξει καλή θέληση η Γαλλία. Τώρα, ποιο θα ήταν το αρνητικό σενάριο, αν δεν δείξει την καλή θέληση η Γαλλία. Το αρνητικό σενάριο θα ήταν να ψηφίσουμε την, την αρχική πρόταση, δηλαδή χωρίς ε, κατεξοδότηση πράξη, αυτό που θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε έτσι θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ανάγνωση με ταπεινοφροσύνη αλλά και με πυγμή και αποφασιστικότητα σας απευθύνω θερμή έκκληση να σταματήσετε το μπλοκάρισμα και να άρετε το βέτο σας ώστε να εξοδετερωθεί αυτή η ανασχετική μειοψηφία συγγνώμη, στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ συνάδελφοι και σας, θα σας θέρμο παρακαλέσω να ε, μείνετε στο ένα λεπτό καθένας. Κυρία Σίπελ. Θα προσπαθήσω. Θα μιλήσω γερμανικά. Κύριε Υπουργέ, είπατε, ε, μιλήσατε για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. έκτακτη ανάγκη όμως έχουμε μόνο όταν τα πράγματα πραγματικά είναι έκτακτα. Οι περιστάσεις είναι εξαιρετικές. Ε, στη Γαλλία, ωστόσο, ε, η κατάσταση αυτή ε, διαρκεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχετε σκοπό να άρετε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ταυτόχρονα είπατε ότι ε, οι ενέργειές σας οδήγησαν στη σύλληψη ε, τρομοκρατών. Μπορείτε να μας πείτε πόσοι ακριβώς έχουν συλληφθεί έπειτα από την ε, κήρυξη κατάσταση έκταξης ανάγκης, πόσοι απελευθερώθηκαν και πόσοι ε, πράγματι καταδικάστηκαν για τρομοκρατικές ενέργειες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το ερώτημα για να δούμε και ποια είναι η επιτυχία των ενεργειών σας. Όσον αφορά τα όπλα, θα ήθελα να μας πείτε τι είδους όπλα αποκαλύφθηκαν και ποιος ο αριθμός τους. Με Μπέρδεψαν λίγο οι αναφορές σας στην Frontex. Συμφωνούμε όλοι ότι τα σύνορά μας πρέπει να ελέγχονται. Ωστόσο, έχουμε και στοιχεία ότι μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό ο νέος ε, οργανισμός ε, της Frontex για την ακτοφυλακή και τη συνοριοφυλακή να αποκτήσει το ε, επαρκές προσωπικό προκειμένου να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του. Τα κράτη-μέλη για, τα, για τους συνοριακούς ελέγχους στην Ελλάδα πρέπει να συμβάλλουν και δεν το έχουν κάνει όλα. Από αυτή την άποψη το ερώτημά μου είναι τι ακριβώς ε, αναμένεται από αυτόν τον ελιγμό. Ίσως ήταν κάποιο πρόβλημα με τη μετάφραση, αλλά τι εννοείται ακριβώς με τον ελιγμό της Frontex. Τελευταίο ερώτημα για το καλέ. Είναι θετικό βεβαίως το γεγονός ότι διαλύθηκε ο καταβλισμός αυτός. Είπατε κι εσείς ο ίδιος ότι ο καταβλισμός αυτός υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Θα ήταν πολύ χρήσιμο φυσικά να είχατε αναλάβει δράση νωρίτερα και να φροντίσετε τους ανθρώπους αυτούς και να μην τους αφήνετε να, στον ισχυρισμό τους ότι θέλουν να πάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, ε, το ερώτημά μου είναι υπάρχουν τώρα πρόσθετες εγκαταστάσεις φιλοξενίας και έχετε αναλάβει μέτρα προκειμένου να αποφύγετε την εκ νέου δημιουργία ενός άλλου καταβλισμού. Επίσης, έχετε στενότερες επαφές με το Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον για τους ανθρώπους εκείνους που πρόκειται να επανενωθούν με τις οικογένειές ώστε να απαστέλλονται αυτοί οι άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Σεσίλια Βίξτρομ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας ε, καλωσορίζω κύριε Υπουργέ. Ήσασταν πολύ δραστήριος όσον αφορά την ανταπόκριση στις ανάγκες ασφάλειας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα στην Γαλλία. Η Γαλλία πίεσε ναι, για την έγκριση, ε, ταχεία έγκριση ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, Ακόμη και αν η ομάδα μου πολλές φορές έχει εκφράσει ανησυχίες ή αμφιβολίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών, παρόλα αυτά, ε, ε, όπως είπατε και εσείς, η κρίση μετανάστευσης είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί από κοινού και σας ακούω και ως εισηγήτρια για τον κανονισμό του Δουβλίνου. Είπατε πολλά για την πολιτική, για την επιστροφή, την επανεισδοχή και το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών, αλλά όσον αφορά το μηχανισμό αλληλεγγύης που προτείνει η Κομισιόν, το στοιχείο της αλληλεγγύης ε, που είναι ε, ο ε, μηχανισμός αυτόματης μετεγκατάστασης. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σας γνώμη, την ε, γαλλική συνεισφορά και προθυμία να συνυπογράψει μια τέτοια κοινή προσέγγιση. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι η Γαλλία μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι υπάρχει ε, μια πολύ μεγάλη απόσταση απέναντι, ανάμεσα στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα, όπου λίγα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, και στη διατήρηση του χώρου Σέγγεν ε, μιας ανοιχτής ε, περιοχής χωρίς συνοριακούς ελέγχους εσωτερικούς. Η συνάδελφος ε, αναφέρθηκε και εκείνη στις, στους κανόνες έκτακτης ανάγκης που έχετε επιβάλει. Έκτοτε, μόνο τρία, τρεις χώρες του μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, παρεκκλίνουν από τις ε, υποχρεώσεις τους με βάση τα, τις συνθήκες που έχουν υπογράψει. Είναι συγκεκριμένα η Τουρκία, η Ουκρανία και η Γαλλία. Είναι αξιοσημείωτο αυτό. Το είπατε, αλλά δεν έχετε απαντήσει στο βασικό ερώτημα που ε, σχετίζεται με, το, με τις αρχές του κράτους δικαίου και την απουσία πρώτερης εκ των προτέρων δικαστικής εντολής για ενέργειες της αστυνομίας. Τέλος, ακούμε ειδήσει σχετικά με τη σύνθεση της γαλλικής κυβέρνησης τις επόμενες μέρες και εγώ ε, σας εύχομαι κάθε επιτυχία και κάθε τύχη ό,τι και αν συμβεί με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ό,τι και να συμβεί, ε, καλό είναι να μην μιλούμε ο καθένας τρία λεπτά, γιατί αλλιώς δεν θα έχει χρόνο ο Υπουργός να απαντήσει. Κύριε ε, κύριε Υπουργέ, καλημέρα και σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Θα, θα ήθελα να συγκεντρωθώ στο θέμα της μετανάστευσης. Να υπενθυμίσω ότι η Γαλλία δεν επλήγει πραγματικά, διότι μόνο κάποιοι χιλιάδες, κάποιες χιλιάδες ετούντες άσυλο ε, μετρήθηκαν το 2015 και υπήρχε σχετικοποίηση με το 2014 και μειώθηκε ο αριθμός τους. Και δέχεται δίνει δικαιώματα, λιγότερο δικαίωμα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι στις έξι χώρες που βρίσκονται στο 30% και πιο κάτω από το 30% όσον αφορά τη χορήγηση ασύλου. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εκτιμήσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλε η Γαλλία για μετεγκατάσταση. Να διευκρινίσω ότι όσον αφορά τον επαναπαντρισμό, η Γαλλία, κατά την άποψή μου, δυστυχώ είναι ένα παράδειγμα. Όλοι οι αριθμοί που έχουμε τη συνήθεια να παραθέτουμε καλύτερο θα ήταν να τίθενται στο κατάλληλο πλαίσιο σε σχέση με τον πληθυσμό μιας χώρας. Η Γαλλία είναι μια από τις χώρες τη πιο πολυπληθής πυκνοκατοικία, μάλλον με το μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ευρώπη και σε σύγκριση με τον πληθυσμό θα στο που καταβάλει με την αντικατάσταση. Για την κατάσταση στο καλέ δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία σας κύριε Υπουργέ. Και ακόμα και την βάση τη επιστολή μου στείλατε 25 Οκτωβρίου όσον αφορά τα ανήλικα παιδιά. Πολλές υποσχέσεις έχουν δοθεί, κυρίως όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση, αλλά οι περισσότερες υποσχέσεις δεν φαίνεται τελικά να επιβίωσαν ε, στο ταξίδι που έκαναν ε, μεταξύ Καλέ και ε, στο Χάσο που όσον αφορά την υποδοχή των παιδιών που έχουν μείνει διάσπαρτα. Λοιπόν, Κάποιοι είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν όλη τη διαδικασία τη άσυλου που είχαν υποβάλει αρχικά στο καλέ στα νέα κέντρα που πάνε. Αλλού υπάρχει ένα μπλοκάρισμα στον αφορά την εξακρίβωση να δούμε κατά πόσο ανήκουν στη, στο σύμβαση του Δουβλίνου ή όχι οι υποθέσεις. Και δεν έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά του οι ετούντο. Και ένα παράδειγμα κύριε Υπουργέ που το γνωρίζετε. Διότι σα είχα ειδοποιήσει αυτό το θέμα. Λοιπόν, Μπαρκέρ από το Σουδάν Α, λοιπόν, ήταν από μια περιοχή που έχει πληγεί από και εμφύλιο πόλεμο. Και παρά τι ειδοποίησει μα, τι δικέ μα και άλλων βουλευτών και των μεγάλων ΜΚΟ, όπω η Διεθνή Αμνηστία, απελάθη αυτό ο άνθρωπο και πήγε στη χώρα προέλευσή του. Και άλλοι υπήκοοι από το Σουδάν ε, κινδυνεύουν να πάθουν τα ίδια. Όμω παρόλα αυτά η Γαλλία πρέπει να πω ότι έχει και το 2015 καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τέλο, ανησυχώ και την κατάσταση στην κοιλάδα της Ραγόγια όπου πολύ πολλά παιδιά έχουν εγκαταληφθεί και η μόνη απάντηση φαίνεται να είναι να στείλουν στα δικαστήρια ε, τους πολίτες που πάνε για να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Ο κύριος Οχτυφέ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Δεν χρειάζεται να βάλετε κάτω ακουστικά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Αναφερθήκατε σε πληθώρα θεμάτων ε, για το... Έχω αφιολογήσει για την πολιτική ασύλου και επιφυλάξει για την πολιτική σας ε, σε ό,τι αφορά την επιστροφή ασυνόδευτων ε, ε παράτυπων συγγνώμη μεταναστών, τις απόψεις για την οδηγία για τα αυτόματα όπλα, αλλά συμφωνώ για τις απόψεις ό,τι αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Εγώ θα σταθώ σε ένα από τα θέματα αυτά για να μην ξεπεράσω τον όρο, το χρόνο που έχω και να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Να αποδείξουμε ότι η Γαλλία μπορεί να δώσει και καλό παράδειγμα μερικέ φορέ. Για το πρώτο ζήτημα τη τρομοκρατία. Ποιο είναι ο αριθμό των τρομοκρατικών επιθέσεων που καταφέρατε να εξουδετερώσετε τον περασμένο χρόνο στη Γαλλία. Επίσης, ποιε απόπειρε επιστροφής μαχητών από τη Συρία και το Ιράκ ε, έχετε αναχαιτήσει την προσπάθεια να επιστρέψουν στο, στη Γαλλική επικράτεια. Πρόσφατα η Ιντερπολ επισήμανε ότι η ομάδα των Σύρων προσφύγων μπορεί να έχει στους κόλπους της και κάποιους ε, ε, τρομοκράτες που έχουν διεισδύσει. Τι γνώμη έχετε γι' αυτό και επίση, πολύ σωστά αναφερθήκατε στο PNR, στο Μητρό Στοιχείων Επιβατών, που προκάλεσε πολλές συζητήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μάλιστα, ο γαλλικό τύπο, πρόσφατα ε, επισήμανε την καθυστέρηση που σημειώνουμε στην εφαρμογή του PNR στη Γαλλία σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο που το εφάρμοσε άμεσα. Έχετε κάποιες εξηγήσει ε, να μας δώσετε για αυτή την ολιγορία που αποβαίνει βάρος του συνόλου του της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μηχανισμού PNR. Ο κύριος Δεπρέ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Έχω μερικές ερωτήσεις ε, για το PNR. Συμφωνώ. Ε, στενίζω με την ερώτηση του κυρίου Ορτφέ. Έχει ε, εφαρμόσει επιτέλους η Γαλλία το μηχανισμό PNR. Μόνο τρεις χώρες φαίνεται ότι έχουν εφαρμόσει αυτό το μηχανισμό μέχρι στιγμής. Ε, κρίμα να έχουμε τέτοιες καθυστερήσεις. Δεύτερον, κλείνει το μικρόφωνο δυστυχώ. σε ό,τι αφορά το άρθρο 7 του κώδικα Σέγγεν, είστε υπέρ των συστηματικών ελέγχων. Ο μηχανισμός όμως που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή προβλέπει τη δυνατότητα απόκληση από τους ελέγχους αυτούς για ένα εξάμεινο ε, που μπορεί να παραταθεί μέχρι τους 18 μήνες ε, εξαίρεση από τους συστηματικούς ελέγχους 6 έως 18 μήνες ανάλογα με ε, την κίνηση. Είναι κάπως περίεργο αυτό. Δεν υπάρχει ένα σοβαρό κριτήριο ασφάλειας, παρά μόνο η ένταση της κυκλοφορίας. επιτρέψτε μου και μία μικρή κριτική προς την ε, γαλλική κυβέρνηση. Αναφέρεται ότι οι ταυτότητες είναι από τα πλέον παραποιημένα έγγραφα και μάλιστα δεν έχουν κάνει ηλεκτρονικό τσίπ ε, οι γαλλικές ταυτότητες. πως κάνω λάθος. Θα είναι δυνατό μια τόσο ελπιμένη χώρα να έχει ταυτότητε που δεν θα είναι τελευταίε γενιέ και δεν έχει καν ηλεκτρονικό τσίπ, να μην έχετε καν ηλεκτρονικό τσίπ στι κάρτε ταυτότητε, στι ταυτότητε γαλλικέ. Ε, για τα ημιαυτόματα όπλα. Θα πρέπει να μα αποδείξετε ότι οι τρομοκράτε έχουν χρησιμοποιήσει τέτοια ημιαυτόματα όπλα. Δεν έχουμε τέτοιε αποδείξει. Η πλειοψηφία των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν από τους τρομοκράτες ε, είχαν αγοραστεί στη μαύρη αγορά. Χρειαζόμαστε τεκμήρια λοιπόν, αποδείξεις αν θέλετε να λάβουμε κάποιες αποφάσεις ε, ε, για να μην ε, λαμβάνουμε απλώς δημοφιλείς αποφάσεις όμως που δεν έχουν αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικές μόνο και μόνο για να γίνουμε αρεστοί στην κοινή γνώμη. Ευχαριστώ. Κύριε Γκόμες. Κύριε Υπουργέ, έχω, έχει την αλληλεγγύη μου, αλλά πάνω σε αυτά που είπατε δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά μιλήσατε για το PNR πτήσεις charter, ευρωπαϊκές πτήσεις είπατε, και ιδιωτικέ πτήσεις σε ένα αεροδρόμιο που είναι τις Νίκες, στο Κασκάι, στην Πορτογαλία Φερρυπίν. Γίνεται έλεγχο των ιδιωτικών πτήσεων που έρχονται με πριγκίψεις στο Ψαδική Αραβία όπως αυτή που, στο, που συνελήφθη ε, με, στο Λίβανο με ναρκωτικά που καταναλώνει η Ντάες συμφωνώ όσον αφορά αυτά που είπατε για τα όπλα και την πέμπτη οδηγία για την οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία όμως. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, περισσότερα δεδομένα, διότι αυτά που έχουμε είναι λίγα. Όπως για τις προπληρωμένες κάρτες, εξασφάλιση, αύξηση ασφαλείας στα σύνορα. Τα κράτη-μέλη μας ασχολούνται με την ενίσχυση συνόρων όσον αφορά τους φτωχούς πρόσφυγες και, τους, και για τους πλούσιους δίνουν χρυσές βίζες και μέσω επενδύσεων. Ποιοι είναι οι διεφθαρμένοι άλλων χωρών που πήραν, ε, πέτυχαν αυτή τη λύση και πήραν θεώρηση μέσω χρημάτων και ποσών στα διάφορα κράτη-μέλη. Εκεί πρέπει να γίνει κίνηση να καταπολεμήσουμε την εγκληματικότητα, αν δεν υπάρχουν ασφαλέ δίωδοι για τους μετανάστες και για τους προσφυγέ. Μήπω τροφοδοτούμε εμείς το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών. Όταν δεν ασχολούμαστε με τα συνότητα παιδιά, δεν δίνουμε ε, ανθρώπους να από τους τρομοκράτες. Όταν δεν ασχολούμεθα με τα παιδιά που βρίσκονται στα στρατόπεδα ε, αυτά τους καταβλισμούς των προσφύγων σε φρικτές συνθήκες όπως στην Ελλάδα. Και τι κάνουμε για την αποφυγή της ασυστοκοπήσης. Υπάρχει πρόγραμμα στη Γαλλία και σε άλλες χώρες για να επιτεθούμε κατά της ριζοσπαστικοποίησης, στις φυλακές, στα προγράμματα ένταξης. Δεν ξέρω τίποτα να υπάρχει πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ Άννα. Κύριε Υπουργέ, το θέμα των πτήσεων τσάρτερ. Θέλαμε να συμπεριλαμβάνονται αυτές το Συμβούλιο ήθελε απλώς σαν ε, επιδυνητικής βάσης. Το αναφέρω αυτό για λόγους ασφαλείας, ότι εμείς το είχαμε αναφέρει, το είχαμε ζητήσει. Η κυρία Ιντεφέλτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Είμαι η Σοφίντ Φέλτ και σύμφωνα με τα γαλλικά με» Σα ταλαιπωρώ. Λοιπόν, πολλέ ερωτήσει ετέθησαν στον αφορά το PNR. Εξεπλάγει, διότι μετά τι πιέσει από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τη στιγμή που ψηφίσαμε φαίνεται, μας πιέσατε να πάρουμε απόφαση, ε, θεωρεί το επίγον, αλλά έκτοτε δεν κινείται τίποτε. Φαίνεται δεν είναι πλέον επίγον. Μετά. Ήξεραν όλοι τότε ότι το πραγματικό πρόβλημα δεν ήταν έλλειψη προσωπικών στοιχείων, το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπάρχει ανταλλαγή των πληροφοριών. Και μέχρι σήμερα εδώ έγκυται το μεγάλο πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω περισσότερα επ' αυτού. Τι γίνεται στο Συμβούλιο. Ασκείται εξίσου πιέσεις στα άλλα κράτη-μέλη για την βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και κυρίως να είναι υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών. Κάτι που είχε ζητήσει η ομάδα μου. Πρώτη τελευταία ερώτηση. Σίγουρα θα μάθατε για την φυγή 700 ε, σελίδες με προσωπικά στοιχεία από έρευνες από την Europol για αντιτρομοκρατικές έρευνες διέρευσαν από την Europol. Το ήξεραν αυτό τα κράτη-μέλη επί σειρά ετών και δεν θα Έπρεπε να το συζητήσουμε και στο Κοινοβούλιο. κυρίως όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών. Και τέλος, είσαστε υπέρ των δημοσίων ελευθεριών. Η κυβέρνηση η γαλλική και η Γαλλία θα προωθεί συζητήσει με το Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά το σύμφωνο, η δημοκρατία, το κάτω δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό που υιοθετήσαμε εδώ και κάποιους μήνες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον τομέα αυτό μαζί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Ζολή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον Υπουργό Εσωτερικών που ήρθε στη συνεδρίαση για να μας παρουσιάσει τις απόψεις του. Στις 30 ε, Οκτωβρίου αποφασίσατε να δημιουργήσετε ένα μέγα μητρό, το ΤΕΣ, στο οποίο περιλαμβάνεται τα δακτυλικά αποτυπώματα και τις φωτογραφίες όλων των Γάλλων, δηλαδή δεκάδες εκατομμυρίων ανθρώπων, δεν πιστεύετε ότι αυτό το διάταγμα που υιοθετήσατε παραβιάζει τους κανονισμούς και ε, τις ε, νομοθετικές διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων που επιτάσσουν την αναλογικότητα, την αναγκαιότητα ως βασικά κριτήρια ε, και για την καταπολέμηση της απάτης υπάρχουν πολύ ε, πιο απλές λύσεις. Όπως ε, το ηλεκτρονικό τσίπ που μπορούμε να συμπεριλάβουμε στην, ε, στην ταυτότητα. Τα εξετάσατε όλα αυτά πριν θεσπίσετε αυτό το μέγα μητρό. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι ως Γαλλίδα νιώθω δυσφορία που ο Ερντογκάν επικαλείται την κήρυξη της γαλλικής ε, κατάστασης ανάγκης για να δικαιολογήσει τη δική του κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ποια είναι τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σουίμπερν. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ναι, ζούμε σε έναν κόσμο όπου φοβόμαστε για την διάπραξη νέων τρομοκρατικών επιθέσεων. Δεν ήταν αυτό το υπόβαθρο όταν αποφασίζαμε την ελεύθερη διακίνηση και τον ανοιχτό χαρακτήρα της Ένωσής μας. Δυστυχώς όμως τα πράγματα ήρθαν έτσι. Ε, εγώ πρέπει να σας ομολογήσω ότι στη Γαλλία ε, αισθάνομαι πολύ πιο ε, ασφαλής από τις άλλες χώρες ακριβώς γιατί έχει, βρίσκεται σε ένα υψηλότερο επίπεδο συναγερμού και χαίρομαι πολύ για τη σύλληψη των επτά αυτών ατόμων που επρόκειτο να διαπράξουν ή σχεδίαζαν να, ε, διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις στο Στρασβούργο. Ε, για τις ε, επιθέσεις ε, είπατε για, τα όπλα, αν και εγώ ε, πρέπει να σας πω ότι σε, αυτές, σε αυτού του είδους τις επιθέσεις ε, δεν γίνεται χρήση καραμπίνων. Ε, νομίζω ότι αυτά τα μέτρα σας στην ουσία πλήττουν τους καημένους κυνηγούς χωρίς κάποια τα αποτελέσματα. Για το καλέ. Καλώς διαλύθηκε ο καταβλισμός, α, όμως το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ε, και εμφανίζονται διαρκώς νέα καλέ σε διάφορα σημεία ε, της ε, Γαλλίας. Ε, επεστράφησαν κάποια άτομα, για παράδειγμα, στην Ιταλία, τα οποία όμως προσπαθούν διαρκώς να ξαναπεράσουν τα σύνορα και να ξαναμπούν στη Γαλλία. Το ερώτημα μου είναι ποια είναι η συνεργασία σας με την Ιταλία όσον αφορά αυτή την επιστροφή. Γιατί τα άτομα αυτά, όπως είπα, επανέρχονται διαρκώς για την ριζοσπαστικοποίηση. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνετε στη Γαλλία. Ελπίζω όμως ότι έχετε θέσει σε ισχύ μέτρα αποτρεπτικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Δύο ομιλητές, πολύ σύντομα όμως παρακαλώ, γιατί ο Υπουργό δεν έχει πολύ χρόνο. κύριος Λιμπρέτο και μετά ο κύριος Στίβενς όσο το δυνατόν συντομότερα, παρακαλώ. Oui, non. Je ne suis pas Monsieur Le Breton, je suis ε, δεν ε, ονομάζομαι Le αλλά Edouard Ferrand. Κύριε Υπουργέ, η Γαλλία ε, συμμετείχε στην, στον πόλεμο στη Λιβύη και στη Συρία. Εσείς δημιουργήσατε το μεταναστευτικό πρόβλημα. Η αποτυχία όμως είναι και ευρωπαϊκή. PNR, ακτοφυλακή, συνοριοφυλακή, Σέγγεν, όλα αυτά τα μέτρα δεν κατάφεραν να εμποδίσουν τους ε, ε, τρομοκράτες Ισλαμιστές να διεισδύσουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δράσουν στην ε, Γαλλία και αλλού. Για τους ε, υπόλοιπους ε, τρομοκράτες λάβατε μεν μέτρα, αλλά ήταν απόλυτα αναποτελεσματικά και στη Γαλλία και στην Ευρώπη γενικώ. Και γι' αυτό κάποιες χώρες επανέφεραν τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και μάλιστα σημαντικές χώρες και γειτονικές χώρες και σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Σήμερα συνεχίζουμε την ίδια άγουσα ε, με πιθανότητα τον επόμενο Φεβρουάριο να απελευθερώσουμε και τις θεωρήσεις προς την Τουρκία. 80 εκατομμύρια Τούρκοι με, τις, με τα σύνορα που γνωρίζουμε, τη Συρία, το Ιράκ, το Ιράν, και τελευταία, τελευταίο σχόλιο για τα όπλα. Εγώ είμαι κυνηγό και πιστεύω ότι θα πρέπει να αφήσουμε την πολυμορφία να λειτουργήσει και εκεί που η κοινή γεωργική πολιτική έχει καταστρέψει το τοπίο μα, ε, να αφήσουμε του κυνηγού ελεύθερου. Πρόκειται για ένα σπόρα. Θα πρέπει λοιπόν να το αφήσουμε ήσυχο. Α μείνουμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, να μην αλλάξουμε τίποτα. Δεν θέλετε να φύγετε από το χώρο Σέγγεν. Πολύ χειρότερα μάλιστα. Θέλετε να ενισχύσετε το χώρο Σέγγεν και πιστεύω ότι θα πρέπει να παραδεχτείτε την πραγματικότητα και γι' αυτό θα ήθελα να σας θέσω μία και μόνο ερώτηση. Πότε θέλετε επιτέλους, πότε θα ακούσετε επιτέλους το μοναδικό αίτημα του λαού που είναι να επαναφέρει την ασφάλεια στα γαλλικά σύνορα. Η κυρία Στίβενς είναι η τελευταία μας ομιλήτρια. Παρακαλώ χρόνου φίδου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που ήρθατε για να συνομιλήσουμε. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις. Πώς πιστεύετε ότι η διάλυση της ζούγκλας του Καλέ, του καταβλισμού του Καλέ ε, θα λειτουργήσει και μπορούμε να κλείσουμε κάποια διδάγματα από την επιχείρηση αυτή της διάλυσης του καταβλισμού. Θέλετε να επαναλάβω την ερώτησή μου. Δεύτερον, η Γαλλίδα αντιμετωπίζει όχι μόνο τη μεταναστευτική κρίση, αλλά και ισχυρότατη τρομοκρατική απειλή. Η Europol συμμετέχει στην Task Force ε, Fraternité, αδελφότητα, που ε, εγκαινιάστηκε μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι το 2015, προκειμένου να ε, στηρίξει τις έρευνες τις βελγο η Task Force έχει αποδείξει μεγάλη αποτελεσματικότητα χάρη και στις πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Και μάλιστα είχαμε ε, τεράστιο όγκο πληροφοριών που, έχει, που έχουν μεταβιβαστεί με αποτέλεσμα να ε, εξουδετερωθούν και κάποιε τρομοκρατικέ ενέργειε. Ποια είναι η εμπειρία σα από αυτό και πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία αυτή τη Task Force. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Είναι πολλέ ερωτήσει. Ευχαριστώ που τι ακούσατε. Έχουμε κάποια λεπτά να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προσπαθήσω δύσκολο να απαντήσω όλε τις ερωτήσεις βέβαια. Θα, δεν έχω τόσο χρόνο στη διάθεσή μου. Δεν θέλω να παραμείνω και παραπάνω από ό,τι πρέπει για να μην υποφέρετε την ε, παρουσία μου. Λοιπόν, θα μπω στο σιώδη λόγω αλληλεγγύων υποχρεώσεων. Για τα υπόλοιπα θα απαντήσω, αν συμφωνείτε, γραπτό να απαντήσω. Θα στείλω τι απαντήσει στον πρόεδρό σα που θα διανύμει τι απαντήσει. Θα προσπαθήσω όμω να είμαι όσο πιο εξεκριτικό γίνεται. Θα ήθελα λοιπόν καταρχά να απαντήσω στο ερώτημα του κ. Διαζεμέρα και να πω ποια είναι η θέση μου, η θέση τη Γαλλία όσον αφορά την απελευθέρωση τη βίζα για τη Γαλλία και τη διαφύλαξη. Να καταλάβουμε ότι η Γαλλία δεν μπλοκάρει Απλώς μέσω της θέσεως που υπερασπιζόμαστε μαζί με άλλους, θέλουμε να είμαστε σε μια θέση ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης να εφαρμόζουμε τις αρχές Ευρωπαϊκής όσο από τη μια, αλλά σε ένα πλαίσιο από την άλλη που λαμβάνει υπόψη ε, τους κινδύνους ε, που είναι συνδεδεμένη με την απελευθέρωση από τις θεωρήσεις αν δεν υπάρχει κάποια ρήτρα διαφύλαξης, αν δεν υπάρχουν μέτρα προφύλαξης, αν δεν υπάρχουν αρχές ή μηχανισμοί που θα μπορούμε να εφαρμόσουμε εάν χρειαστεί κάποια δεδομένη στιγμή. Αν γίνει ανεξέλεγκτη η κατάσταση, διότι αν δεν είμαστε σε θέση να έχουμε δυνατότητα ρύθμιση στην Ευρώπη, αν η Ευρώπη δεν μπορεί να ελέγξει τις συνέπειες των ηλυμένων αποφάσεων, να μην εκπλήσεστε για την άνοδο του λαϊκισμού. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν αρχές, κανόνες, ρύθμιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε λοιπόν σε διάφορες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση θεωρήσεων, κυρίως με την Τουρκία, τη Γεωργία, την Ουκρανία και το Κωσυφοπαίδιο. Είναι ένα θέμα, έχω επίγνωση αυτού, ε, πάρα πολύ ευαίσθητο πολιτικά και θα πρέπει να προσμετρήσουμε με προσοχή τις συνέπειες των αποφάσεων που θα λάβουμε μαζί. Και το επαναλαμβάνω, πώς εξηγείται συλλογικά, μακροπρόθεσμα και ήδη στην κοινή μας γνώμη ότι σε ένα πλαίσιο απειλής μεγάλης από την τρομοκρατία και μεγάλων μεταστρεπτικών ροών αποφασίζουμε να ανοίξουμε το χώρο μα, ο οποίο είναι πάρα πολύ εύθραυτο ήδη, τη ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων, χωρί να έχουμε δυνατότητα ελέγχου και ε, προστασία. Θα ήταν δύσκολο, δυσνόητο κάτι θα ακούγαμε μεγαλύτερε επικρίσει. Διότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν δίνει ευκαιρίες ελεύθερης διακίνησης δεν προστατεύει ταυτόχρονα, τότε θα υπάρχει μεγάλη απομάκρυνση της κοινή γνώμης από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και ανοίγουμε ανοιχτά τις πόρτες του λαϊκισμού, κάτι που δεν επιθυμεί η Γαλλία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν είναι μόνο η Γαλλία άλλωστε. Ζητήσαμε εμείς από τον Τόμας Δεμεζιέρ, τον ομολογό μας και από άλλες χώρες που είναι ευαίσθητε για αυτό το θέμα, για αυτό το διάβημα που κάνουμε, η διαδικασία τη απελευθερώσεω των θεωρήσεων να είναι καλά πλαισιωμένη. Αποστήλαμε προτάσει ε, τέλο ε, του μήνα Απριλίου προτείνοντα την ύπαρξη μιας, μηχανισμού διαφύλαξη που θα επιτρέπει την αναστολή τη απελευθερώσεω θεωρήσεων υπό κάποιου όρου που είναι ακριβέστατοι. Αυτό ο μηχανισμό δεν είναι μια εφεύρεση τη Γαλλία που θα μπλόκαρε όλα ξαφνικά. Ο μηχανισμό αυτό θεσπίστηκε το 2013 καθορίζει τα κριτήρια που κατά την άποψή μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να πληρούνται και βασίζονται επί διαδικασίας πάρα πολύ άκαμπτης. Δεν εφαρμόστηκε για την απελευθέρωση των θεωρήσεων σε προηγούμενες περιπτώσεις λόγω ακαμψίας και λοιπόν η πρότασή μας έχει σαν στόχο να γίνει πιο εύκαμπτος ο μηχανισμός. Τρεις αρχές οδήγησαν το, το Συμβούλιο συγγνώμη, στην προσέγγιση κριτήρια αντικειμενικά για τη χρήση του μηχανισμού, ταχείας εξέτασης διαδικασία, και τρίτον, να καταλήγουμε σε αναστολή της εξαίσθησης θεωρήσεως όταν τα κριτήρια εφαρμογής του μηχανισμού διαφύλαξης πληρούνται. Το συζητούμε αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη δική σας Επιτροπή, μάλλον συζητήσει στον τριμερή διάλογο με την Επιτροπή σας, οδήγησε σε σημαντικές προόδους. Θα ήθελα να χαιρετήσω το συμβαστικό πνεύμα που επιδείξατε. Θα ήθελα το συμβαστικό πνεύμα που επικρατεί, που είναι και δικό μας συνεργάσιμο πνεύμα, μαζί με άλλες χώρες στο τριμερή διάλογο να οδηγήσει τελικά σε μια θέση που προδεύει. Και ίσως μέχρι τώρα τέλος συζητήσεων, καταλήξουμε σε κοινή θέση, θα είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Λοιπόν, να πω στην κυρία Σίπελ και σε άλλους ευρωβουλευτές που εκφράστηκαν απλά πράγματα όσον αφορά την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και για το καλέ. Όσον αφορά την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν είναι μια παράβαση μονομερής πλευράς του κράτους κινούμεθα στα πλαίσια του δικαίου, το κράτος δικαίου στη Γαλλία. Για, ότι παραβιάσαμε το κράτος δικαίου στη Γαλλία. Δεν είναι παράβαση. Ε, η κατάσταση κατεπηγούσης ανάγκης στη Γαλλία είναι ένας μηχανισμός του 1955, θεσπίστηκε, του γαλλικού δικαίου, που ανανεώθηκε τη στιγμή που έπρεπε να λάβουμε μέτρα την επόμενη ημέρα των, των επιθέσεων του Νοεμβρίου του 2015 και χρονολογείται το 1955 η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης προβλέπεται από το γαλλικό δικαίου. Εν πουδενή δεν λησμονήσαμε και αγνοήσαμε ε, τον νόμο για να κάνουμε πιο αστυνομικό το κράτος ε, μονόπλευρα και αυθαίρετα. Υπάρχει ένας μηχανισμός που προβλέπει το γαλλικό δίκαιο, επιτρέπεται και επιτρέπει στη, στην κυβέρνηση όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος και στη δίκηση και όταν διακηρύσσει την κατάσταση εκτάκτου ανάγκη για να παραταθεί, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι υπάρχει άμεσο κίνδυνο και η διοικητική αστυνομία προστατεύει λοιπόν του Γάλλου από την, με μέτρα, του Γάλλου από την τρομοκρατία. Στα πρέσια σεβασμού του νόμου λαμβάνονται τα μέτρα, ελέγχονται νομικά τα μέτρα και από το Κοινοβούλιο ελέγχονται. Η Επιτροπή του Νόμου της Εθνοσυνελεύσεως και της Γερουσίας, οι αρμόδιες επιτροπές αποφάσισαν να εφαρμόζουν μόνιμα τον έλεγχο της εφαρμογής καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης. Και οι βουλευτές μπορούν να πηγαίνουν σε, όλες, σε όλους τους νομούς της Γαλλίας συνεχώς για να ελέγχουν τις συνθήκες επί τις οποίες οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης. Η επιτροπή αυτή, η κοινοβουλευτική, είναι ισχυρή, ε, λογοδοτεί σε μια ειδική επιτροπή του Κοινοβουλίου και γίνονται κατάλληλε συζητήσει στο Κοινοβούλιο τη Γαλλία. Είναι δυναμικέ, ζωηρέ, ε, όπω και στη δική σα επιτροπή σήμερα οι συζητήσει είναι ζωηρέ και είναι καλό αυτό. Δεν μπορεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκη να γίνεται ε, χωρί τον έλεγχο τον κοινοβουλευτικό. Μετά υπάρχει έλεγχο του δικαστού. Ο διοικητικό δικαστή θα πρέπει να ελέγχεται Καταλαβαίνω ότι εδώ δεν γνωρίζετε όσο η Γάλλοι νομικοί πάντα τις λεπτομέρειες του γαλλικού δικαίου. Στη Γαλλία λοιπόν ο διοικητικός δικαστής ε, είναι ένας δικαστής που ε, φροντίζει για τα θέματα αυτά. Όπως είναι ανεξάρτητος και ασκεί όσον αφορά τις δράσεις αστυνομικής, ε, διοικητικής αστυνομίας ε, την ελέγχει αυστηρά και το Συμβούλιο Επικρατείας. Δεν είναι η αρχή που απαιτεί τους ελέγχους δυνάμει της συνταγματικής αρχής που προβλέπεται και σύμφωνα με τη Γενική Νομοθεσία, οπότε το Συμβούλιο Επικρατείας μπορεί να ε, προβάλλει αντίρρηση να καταρρύψει κάποιες αποφάσεις που δεν είναι σύνομες. Λοιπόν, είναι ένας μηχανισμός που προβλέπεται από το κράτος δικαίου, η κατάσταση εκτάκτη ανάγκης και από τον αρμόδιο δικαστή ελέγχεται. Να πω, ο ίδιος ο δικαστής ε, απαιτεί τίτε να επέμβει σε περίπτωση μέτρων που απορρέουν από την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης όταν αυτό που ανακαλύπτεται σε περίπτωση ε, αυτή επιτρέπει την, την παρέμβαση του δικαστού του ποινικού δικαίου όταν αυτό που αποκαλύπτονται το ζητούν, απαιτούν κάτι τέτοιο και ο δικαστής μπορεί να αποφανθεί όσον αφορά τις διοικητικέ έρευνε ή τι ε, τις διάφορες κατοίκων έρευνες. Όταν ακούω κάποια σχόλια όσον αφορά την κατάσταση εκτάκτου ανάγκη στη Γαλλία και βλέπω ποιο είναι και ένα νομοθεσίσμα από αυτού, βλέπω ότι υπάρχει διαφορά, απόκληση. Καταλαβαίνω ότι στην πολιτική σφαίρα ή στη δημόσια συζήτηση μπορούμε να παρασυρθούμε από τη συζήτηση, να εκφράζουμε και επιθυμίε και να υπάρχουν, θέλουμε, περισσότερου ελέγχου. Αλλά η πραγματικότητα στον αφορά την κατάσταση εκτάκτου ανάγκη στη Γαλλία είναι αυτή. Είναι το κράτο δικαίου, κυρία Βερζιά, που ισχύει. Μπορείτε να με κοιτάτε υπομειδιώντα, αλλά υπάρχουν ε, έχετε δικαίωμα το ρωτάτε. Λοιπόν, το κράτος δικαίου υπάρχει αυτή η νομοθεσία στη Γαλλία και υπάρχει και νομολογία και υπάρχει και το Συμβούλιο Επικρατείας και υπάρχουν οι διάφοροι νόμοι, τα διάφορα πλαίσια, συνταγματικά πλαίσια. Μπορείτε να υποκρίνεστε ότι δεν υπάρχουν αυτά, ε, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε το θέμα με σοβαρότητα και θεωρητική. Δεν μπορώ να σας αφήσω να λέτε ότι κατεπήγουσα η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι η πλήρης αυθαιρεσία. Δεν αληθεύει. Και γι' αυτό λοιπόν προβλέψαμε και μεγάλη παρέμβαση των δικαστικών αρχών και το Κοινοβούλιο κάνει τη δουλειά του επ' αυτού. Με ρωτήσατε για κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν εσείς θέσατε το ερώτημα ή κάποιος άλλος συνάδελφός σας που σωστά με ρώτησε γι' αυτό. Α, η κυρία Σίπελ. Ποια είναι τα αποτελέσματα που πετύχαμε στα πλαίσια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και πόσοι άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Λοιπόν, όσον αφορά τον αριθμό των συλληφθέντων από την αρχή του έτους ε, που θέσατε το ερώτημα αυτό, 418 συλλάβαμε από την αρχή του έτους στη Γαλλία. Αυτό δείχνει το επίπεδο της τρομοκρατικής απειλής που αντιμετωπίζουμε. Να υπενθυμίσω ότι να γίνεται μια απόπειρα στη Γαλλία, ε, το εκτελεστικό κλάδος θα πρέπει η εκτελεστική εξουσία πρέπει να επιληφθεί. Ε, και αυτό είναι η ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο, πολιτική ευθύνη. Και γι' αυτό, λοιπόν, να σας δώσω λοιπόν το επίπεδο της απειλής, να δείτε ποια είναι η ένταση και των δραστηριοτήτων των μυστικών μας υπηρεσιών. 418 συλλήψεις ατόμων που συνδεόταν με τα τρομοκρατικά δίκτυα από τις αρχές του έτους του 2016, από την 1η Σεπτεμβρίου 143 συλλήψεις, 52 μάλλον 21 είναι από τον δικαστικό έλεγχο για το μήνα Νοέμβριο που πέρασε. Οι τρομοκρατικές ομάδες συνέλαβαν 43 ανθρώπους, 28 παρεπέμφθησαν και περίπου 20 σχέδια επιθέσεων ε, ανακαλύφθηκαν και απετράπησαν. Με ρωτήσατε ποιος ήταν ο αντίκτυπος της καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης όσον αφορά τις συλλήψεις. Πραγματοποίησαμε από το μήνα Ιούλιο 543 διοικητικές ερευνές που επέτρεψαν να βρούμε όπλα, όπλα, πολεμικά όπλα, ε, ο, όπως ε, μαχαίρια και άλλου είδους όπλα, όταν ξέρουμε ότι υπάρχει ε, δυνατότητα επαφής μεταξύ των διαφόρων ομάδων, εγκληματικών ομάδων με τους τρομοκράτες, υπάρχει επαφή και πολλοί από αυτούς που είχαν καταδικαστεί για τρομοκρατία προηγουμένως είχαν καταδικαστεί για διάφορα δικήματα και βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Την περασμένη εβδομάδα ε, κάποιο που υπέστη έρευνα συνελήφθη, ε, συνεκεία φυλακίστηκε για σχέσεις που είχε με τρομοκρατική ομάδα. Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι χρήσιμη. Δεν λέω ότι στα πλαίσια της καταστάσεως αυτής δεν κάναμε έρευνε οι οποίε δεν οδήγησαν σε απτά αποτελέσματα σε σχέση με του τεθέντε στόχου. Αυτό θα ήταν ψεύδο, αλλά ήταν χρήσιμη κατάσταση. Αρχέ Νοεμβρίου 2016, 687 άτομα γαλλικής υπηκότητας που διαμένουν στη Γαλλία είχαν σχέση με το φαινόμενο που ανέφερα. Οπότε, όπω καταλαβαίνετε, η κατάσταση εκτάκτου ανάγκη είναι πραγματικά απαραίτητη και χρήσιμη. Μετά με ρωτήσατε για το άλλο θέμα όσον αφορά το Frontex. Και το καθήκον της Γαλλίας ε, για τη Frontex ε, και το Καλέ. Θα σας μιλήσω για αυτά τα τρία και για τη διαδικασία της ε, μεταγκατάστασης. Ό,τι αφορά το Καλέ, κυρία Βερζιά, να σας δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση. Στο Καλέ τους τελευταίους μήνες, από τον Οκτώβριο του 2015 είχαμε 13.000 ε, άτομα που μετακαταστάθηκαν σε θέματα υποδοχής και προσανατολισμού και 2.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι στα πλαίσια των πρόσφατων επιχειρήσεων. Αυτά είναι τα συγκεκριμένα νούμερα. Από τον Οκτώβριο του 2015 και την πρόσφατη επιχείρηση είχαμε 13.000 άνθρωποι που μεταφέρθηκαν σε ε, κέντρα φιλοξενίας και προσανατολισμού, εκ των οποίων 2.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι. Και μάλιστα κοινοποιήσαμε πολλές ε, ενώσεις, ε, γιατί ενώσεις ε, διαχειρίζονται αυτά τα κέντρα υποδοχής φιλοξενίας και προσανατολισμού και σε καμία περίπτωση δεν είναι μήνυ καταβλισμοί προσφύγων αυτά τα κέντρα φιλοξενίας. Πρόκειται για κέντρα δεσπαρμένα στη Γαλλική επικράτεια, που είναι ένας ενδιάμεσος σταθμός μεταξύ της λάσπης, του κρύου, της επισφάλειας, της βίας στο έλεος των ελαθροκινητών και των κέντρων υποδοχής των τον άσυλο στα πλαίσια του εθνικού συστήματος. Μεταξύ των 13.000 που στείλαμε από το Καλέ σε κέντρα προσανατολισμού και φιλοξενίας, 80% αυτών των 13.000 ζήτησαν ε, άσυλο στη Γαλλία. Και όταν ε, ακούω μερικούς συγκεκριμένες ε, ε, πολιτικής ιδεολογίας, αριστερά κυρίως του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που λένε ότι ήταν πολύ χαμηλός ο αριθμός των ετών των άσυλων, 80 με 85% των θαμώνων του Καλέ ζήτησαν άσυλο από τη Γαλλία. Τώρα, όταν ακούω άλλες δεξιάς παράταξης ευαισθησίες που λένε ότι το γεγονός ότι η μεταφορά αυτών των θαμώνων του Καλέ στο Εθνικό Σύστημα Προστασίας Ασύλου ισοδυναμεί με μαζική νομοποίηση ή χορήγηση δικαιωμάτων, ούτε και αυτό αληθεύει, γιατί αυτό που κάναμε στα πλαίσια του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ασύλου ήταν άνθρωποι που ήταν επιλέξιμοι ε, για την ε, προστασία αυτή. Ήταν άνθρωποι που δεν ήταν επιλέξιμοι για απελάσεις. Δεν επρόκειτο να βάλουμε διοχθέτες από τον Πασάρ Ελλάς αντί για ζήτη ε, σε, στο, σύστημα αυτό. και μάλιστα ελάχιστες αποχώρηση είχαμε από τα κέντρα υποδοχής και προσανατολισμού. Στα κέντρα υποδοχής και προσανατολισμού ε, οι άνθρωποι που έφτασαν από το Καλέ ε, ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους. Δεν είναι άνθρωποι που εμπίπτουν στον κανονισμό του Δουβλίνου, γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι ουσιαστικά εντείνουμε την επισφάλεια. Όχι, δεν το κάνουμε. Έγραψα σε πολλές ενό για να δώσω απαντήσει στι απορίε του για το θέμα αυτό και το γεγονό ότι ε, δεν το κάνουμε δεν σημαίνει ότι στα κέντρα υποδοχή και προσανατολισμού δεν εφαρμόζουμε το σύνολο των διαδικασιών που πρέπει να εφαρμοστούν. Γιατί το γεγονό ότι δείχνουμε ανθρωπισμό δεν σημαίνει ότι ξεχνούμε τι αρχέ του δικαίου που πρέπει να ισχύουν σε τέτοιε περιπτώσει. Τώρα, για, τα, για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Επαναλαμβάνω, 13.000 ανθρώπους ε, ε πήραμε από το καλέ. 2.000 από αυτού αυτούς είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Ε, αυτοί ισχυρίζονται ότι είτε έχουν οικογένεια στη Μεγάλη Βρετανία, είτε ε, εμπίπτουν σε μια διάταξη. Ε, πάντως, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που ε, ε σώθηκαν από την επισφάλεια και την λάσπη του Κάλε δεν έπρεπε να πάνε σε κέντρα φιλοξενίας ε, που τις χειρίζονται οι ε, ενώσεις αυτές και η άλλη επιλογή ήταν να τους μεταφέρουμε στην ε, Μεγάλη Βρετανία. Η Γαλλία έκανε τεράστιες προσπάθειες ε, για να βάλει στο Εθνικό Μηχανισμό Ασύλου ανθρώπους που ήταν ευάλωτοι και που δεν θα ζητούσαν το άσυλο στην Γαλλία αλλά στη Μεγάλη Βρετανία. Και εμεί κάναμε την προσπάθεια με το Γαλλικό Γραφείο Μετανάστευσης και τους συμπεριλάβαμε στον Εθνικό Μηχανισμό Ασύλου και θα ήθελα η Γαλλία που έκανε αυτές τις τεράστιες προσπάθειες να μην βρεθεί μόνη της στις προσπάθειες αυτές και να συνοδευτεί η προσπάθεια αυτή από τις αντίστοιχες προσπάθειες άλλων χωρών. Κυρία Σίπελ, κυρία Βεριζιά, θα πρέπει και οι Βρετανοί να συνεχίσουν να κάνουν προσπάθειες και η συνεργασία μας συνεχίζεται. Η Γαλλία ζητάει και από άλλες χώρες να κάνουν προσπάθειες όπως ε, και εμείς, τουλάχιστον, ε, τουλάχιστον ισοδύναμες με τις δικές μας προσπάθειες. Και αυτό θα ήθελε να γίνει με καλές, καλούς όρους και μάλιστα σχετικά γρήγορα. Η Γαλλία ανέλαβε τις ευθύνες της για το καλέ. Και μπορείτε να μου λέτε ό,τι θέλετε, αλλά τα κέντρα φιλοξενίας και ε, προσανατολισμού, όπου πρόσφυγες έχουν βρει τροφή, στέγη, ζεστα, ζέστη, θαλπορή. Είναι πολύ καλύτερα από τη λάσπη και το κρύο του καλέ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να αναλάβει μια χώρα τις ευθύνες της. Μην μου λέτε λοιπόν ότι ενώ είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που έχουν καταφέρει να, διαλύσουν ένα καταβλισμό προσφύγων όχι δια, διαχέοντας και σκορπίζοντας αριστερά και δεξιά τους πρόσφυγες, αλλά προσφέροντάς τους ε, τροφή και στέγη ε, και ζέστη, μη μου λέτε ότι εμείς δεν κάναμε τίποτα. Νομίζω ότι μπορούμε να νιώθουμε υπερήφανοι για τον τρόπο που χειριστήκαμε τη διάλυση του καταβλισμού του Καλέ. Και αν αντιμετωπίσουμε δυσκολίες με κάποιους ε, ευάλωτους, θα, θα εφαρμόζουμε τις αρχές προστασίας που ισχύουν με το σεβασμό των αξιών και των αρχών μας. Τώρα, θα πρέπει και για τη Frontex να κάνουμε το καθήκον μας και εμείς ε, συνεισφέρουμε, είμαστε από τους βασικούς ε, συνεισφορεί ε, στο Frontex. Από τους 1500 έχουμε 170 Γάλλους αποσπασμένους και αν προσθέσουμε τους το προσωπικό, του τους μεθοριοφύλακες που στείλαμε στην Ελλάδα με αίτημα της Ελλάδας, γιατί μερικές φορές οι Έλληνες μόνο τους έχουν να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες δυσκολίες και χρειάζεται να υποδεχθούν και να περιθάλψουν στα κέντρα καταγραφής χιλιάδες πρόσφυγες για να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τους κατάλληλους όρους και συνθήκες. Είναι αδύνατο να το κάνουν χωρίς τη δική μας συνεισφορά. Και μάλιστα η Γαλλία έχει αναλάβει δεσμεύσεις που τηρεί αυστηρότατα και θα συνεχίσει να το κάνει γιατί αυτό είναι ο ρόλος να εκπληρώσει το καθήκον της. Μου είπατε πόσες ε, τρομοκρατικές επιθέσεις εξουδετερώσαμε, αποτρέψαμε. 17 τρομοκρατικές επιθέσεις αποτρέψαμε. Και θα πρέπει να το συνδυάσετε με τον αριθμό των συλληθέντων που σας ανέφερα. Δεν ξέρω αν ε, διανοήσετε τι σημαίνει 418 συλληθέντες ε, και πολλοί μάλιστα έχουν ε, φυλακιστεί για σχέση με τρομοκρατικά δίκτυα ή για υποψίες τρομοκρατικών ενεργειών. Και μάλιστα συλλάβαμε και τρεις νεαρές γυναίκες ε, που σε Αντουάν την ώρα που προσπαθούσαν να επιτεθούν σε έναν αστυνομικό. Γιατί εμείς παρακολουθούσαμε, ξέραμε ότι θα περάσουν από στα έργα και υπήρχε σοβαρότατο κίνδυνο διάπραξη σοβαρού εγκλήματος και μάλιστα στην επιχείρηση της μασαλία και του Στρασβούργου τη περασμένη εβδομάδα, είχαμε την εξάρτηση ενός πυρήνα ε, τύπου της 13ης Νοεμβρίου, των τρομοκρατών τη 13 η Νοεμβρίου που σκόπευαν να κάνουν μαζικέ επιθέσεις ε, επίσης και στο, σε μια συνοικία του Παρισιού εντοπίσαμε ένα πυρήνα με τεράστιο πλωστάσιο που επρόκειτο να οργανώσει επιθέσεις με κρυκτικά δολοφονικές στην Γαλλία. Βλέπετε λοιπόν τι απειλές αντιμετωπίζουμε και προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις ικανότητες των μυστικών μας υπηρεσιών και των, της αστυνομίας να βελτιώσουμε τις συνθήκες κινητοποίησης με αυστηρό σεβασμό των προσωπικών δεδομένων και το, του ευρωπαϊκού δικαίου τις ε, α, τεχνικές α, των μυστικών υπηρεσιών για εντοπισμό τρομοκρατικών ενεργειών και προσπαθούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ του απόλυτου σεβασμού των ελευθεριών και φυσικά είμαστε ρεπουμπλικάνοι και μας είναι προσφυλής αυτή η παράδοση και τις ανάγκες να εξασφαλίσουμε την προστασία των Γάλλων ο αριθμός των ε, τζιχαντιστών που επέστρεψαν. Περίπου 200, 203 συγκεκριμένα. 219 έχασαν τη ζωή τους ε, επί τόπου, κάτι που δείχνει το έβρος αυτού του φαινομένου. Και αν δούμε μόνο τη Γαλλία, 2.000 στη Γαλλία έχουν κάποια σχέση με την τρομοκρατία. 1.100 ε, είχαν μεταβεί στο Ιράκ και τη Συρία και από αυτούς 400 έχουν επιστρέψει, 700 βρίσκονται ακόμη ε, Συρία-Ιράκ και έχουν χάσει τη ζωή τους ε, σε τέτοιες ζώνες. Πρόκειται για ένα φαινόμενο μεγάλων διαστάσεων, ιδιαίτερα ανησυχητικό. Και οι υπόλοιποι χίλιοι είναι άτομα που βρίσκονται στο δρόμο μεταξύ Ιράκ, Συρίας και Γαλλίας. Είτε ήδη βρίσκονται στο έδαφος μας ε, ή ανα πάσα στιγμή μπορούν να εισέλθουν στο εδαφός μας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό και ανησυχητικό φαινόμενο με μεγάλες διαστάσεις και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε ε, γενικές πολιτικές καταπολέμησης τρομοκρατίας ε, και πάταξης της ε, ριζοσπαστικοποίησης. Τώρα, για την απορριζοσπαστικοποίηση. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και προσπάθειες που κάνουμε απορριζοσπαστικοποίησης και στη Γαλλία και στην Ευρώπη. Και στη Γαλλία έχουμε ε, καλύτερη οργάνωση της επικοινωνίας μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών και αυτή τη στιγμή 5.000 νέοι έχουν εντοπιστεί στην σχετική πλατφόρμα που εμπίπτουν στη διαδικασία απόρριζος παστικοποίησης ε, υπό την επιτήρηση των εισαγγελέων κινητοποιώντα τι τοπικέ κοινότητε και ειδικευμένε οργανώσει που συμβάλλουν σε αυτή την απορριζοσπαστικοποίηση, με κέντρα απορριζοσπαστικοποίηση και μάλιστα έχουμε στενή συνεργασία και με κάποιους φορείς στο ίντερνετ ε, για να αναπτύξουμε ένα εναλλακτικό αφήγημα και να εντοπίσουμε κάποιες ε, ιστοσελίδες που προωθούν, εκθιάζουν την τρομοκρατία και ήμασταν η πρώτη χώρα που συνήψε σύμβαση με ε, παρόχους υπηρεσιών στο ίντερνετ για να μπορέσουμε να κλείνουμε σελίδες στο ίντερνετ. Έχουμε μεγάλη πρόοδο και στο θέμα της απόσυρσης σχετικών ιστοσελίδων. Επίσης, έχουμε κινητοποιήσει φορείς της κοινωνίας των πολιτών για να παρουσιάσουμε μια εναλλακτική ε, αντιτρομοκρατική ρητορική και έχουμε και ένα δίκτυο που έχει εξέπαινο έργο στο θέμα της απορριζοσπαστικοποίησης. Έχουμε τεράστιες λοιπόν πρωτοβουλίες ε, υπέρ της απορριζοσπαστικοποίησης, πολύ θετικές. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση της κυρίας Ζολή, για το Μητρό ΤΕΣ. Είπατε ότι το Μητρό αυτό αντιβαίνει στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Καταρχήν αυτό το Μητρό ε, υπάρχει, υπάρχουν δύο Μητρό, το Μητρό ΤΕΣ που αφορά 30 εκατομμύρια Γάλλους ε, για τα βιομετρικά όσοι έχουν βιομετρικά διαβατήρια και έχουμε και το Εθνικό Μητρό Διαχείρισης που περιλαμβάνει ήδη τα δακτυλικά αποτυπώματα 60 ε, εκατομμύριων Γάλλων. Δεν ήταν ψηφιοποιημένο, ήταν ε, σε χαρτί ε, με λιγότερη χνηλασιμότητα από το Μητρό ΤΕΣ. Πάντως, το Μητρό ΤΕΣ Έχουμε ήδη νομολογία το Απριλίου 2015 για την ε, εθνική ταυτότητα και, και το Γαλλικό Συμβούλιο Επικρατείας εξέτασε τη συνταγματικότητα αυτού του διατάγματος, ώστε το ε, αρχείο το μητρό τεστ που χρησιμοποιείται για τα διαβατήρια να επεκταθεί και στις ταυτότητες. Και αν ε, η, Ευρωπαϊκή Αρχή για τις Ελευθερίες ε, έχει εκφέρει κάποιες αφιβολίες σε καμία περίπτωση δεν ε, είπε ότι είναι παράνομη αυτή η διαδικασία. Ούτε αναφέρθηκε ουδέποτε ότι οι ενέργειές μας ε, ήταν αντισυνταγματικές ήταν παράνομες. Οπότε, από αυτήν την άποψη, έχουμε το πράσινο φως από το δικαστήριο για το εγχείρημα. Αυτό που είπε όμως η αρμόδια αρχή για τις ελευθερίες είναι ότι Δεδομένη της σημασία του θέματος έπρεπε να γίνει ε, κοινοβουλευτική συζήτηση. Θα συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή μετά τις αιτήσει που έγιναν στην ε, Εθνική Αρχή Ασφάλειας και είπαμε ότι από τη στιγμή που δεν ήταν δυνατόν να προχωρήσουμε στο μετρό με τον εντοπισμό με βάση τα βιομετρικά στοιχεία αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εντοπισμό της ταυτότητας, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η αντιστρεψιμότητα του μηχανισμού δεν θα ήταν δυνατή, ώστε να γίνει απόλυτο σεβασμό στις προστασίες των δεδομένων. Ζήτησα περαιτέρω διερεύνηση του θέματος από τους ειδικευμένους φορείς της Γαλλίας ώστε να εξασφαλιστούν όλα τα εχέγγυα για το θέμα αυτό και είπα, δεσμεύτηκα ότι θα δημοσιεύσω όλες αυτές τις έρευνες ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την θέλησή μας να βελτιώσουμε την ασφάλεια των στοιχείων της ταυτότητας χωρίς να διακυβεύουμε τις προσωπικές ελευθερίες. Επίσης, ένας συνάδελφός σα μας μίλησε για την ύπαρξη ηλεκτρονικού τσίπ στα, στις ταυτότητες ε, για έναν απλούστατο λόγο δεν διαλέξαμε αυτό το σύστημα. Εμείς ε, θέλησαμε να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα στους Γάλλους να ανανεώνουν αμέσω ε, την ταυτότητά τους, χωρίς να χρειάζεται να επαναλάβουν όλες τις διατυπώσεις που θα έπρεπε να κάνουν αν είχαν τσίπ ε, ηλεκτρονικό στο εθνικό δελτίο Ταυτότητες. Για απλούστευση της διαδικασίας λοιπόν δεν υιοθετήσαμε αυτό το τσίπ και αυτή, αυτός ήταν ο λόγος που κάναμε τη συγκεκριμένη επιλογή και μάλιστα το εξήγησα αυτό και στη Γαλλική Εθροσυνέλευση όπου παρήχα και όλες τις πληροφορίες σχετικά. Αυτά δεν μπόρεσα δυστυχώς να καλύψω όλα τα θέματα και λυπούμε, αλλά δυστυχώς πρέπει να φύγω, έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις, πάντως σας υπόσχομαι να σας στείλω γραπτός απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που δεν πρόλαβα να καλύψω. Α, συγγνώμη. Θα ήθελα οπωσδήποτε να ε, δώσω την απάντηση για το Σέγγεν, PNR λοιπά. Η ομάδα έχει μια πολύ κλασική θέση για το θέμα αυτό. Ψηφίστε συστηματικά κατά όλων των ε, προτάσεων και στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είστε κατά του PNR, ήσασταν κατά των, της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας ε, που καταθέσαμε στη Γαλλία. Υπάρχει μόνο μία λύση, την επαναφορά του ελέγχου στα σύνορα. Ε, βέβαια, δεν θα πρέπει να διαφεύγει τη οξυδέρκειά ότι ε, ο έλεγχο στα σύνορα επανήλθε από τι 13 ε, Νοεμβρίου του 2015 και ότι ισχύει αυτό ο έλεγχο. Και μάλιστα έχουμε διασφαλίσει ε, την προστασία των σύνορων χάρη στην επαναφορά αυτών των ελέγχων. Και μάλιστα είμαστε στην αιχμή τη μεταρρύθμιση του Σέγγεν προκειμένου να ενισχυθεί και η Frontex, να γίνονται αποτελεσματικοί έλεγχοι στα σύνορα και χάρη σε συστηματικό έλεγχο και του συστήματος Σέγγεν Προσπαθούμε και στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδυάσουμε το Μητρό Σέγγεν με άλλα Μητρώα ε, με τη Eurodac και τον αναθεωρημένο ε, κανονισμό ε, είπαμε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λόγους εσωτερικής ασφάλειας και μάλιστα η Γαλλία έχει μια θέση σε ό,τι αφορά τους ελέγχους στα σύνορα και η τροφοδότηση του συστήματος πληροφοριών του Σέγγεν από τις μυστικές υπηρεσίες ή συστηματική, ο συστηματικός έλεγχος του συστήματος πληροφορικής του Σέγγεν, ο συνδυασμός του συστήματος Σέγγεν με άλλα μητρώα του ποινικού δικαίου. Ο αντιτρομοκρατικός αγώνας βρίσκεται στο επίκεντρο όλων αυτών των προσπαθειών. Και για όλα αυτά τα θέματα η Γαλλία βρίσκεται στην αιχμή και αναλαμβάνει όλες τις πρωτοβουλίες και δεν πρόκειται με τη δημαγωγία να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την τρομοκρατία. Σας ευχαριστώ. Υπουργέ, πρωτού φύγετε να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της Επιτροπής. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση. Δεν έρχονται πολλοί ε, συχνά υπουργοί από τις μεγάλες χώρες ε, στις συνεδριάσεις μας. Το έχετε κάνει επανειλημμένο και ξέρω και, και πρέπει να σας πω ότι το εκτιμούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά τα θέματα και πολύ ενδιαφέροντα για το PNR και όλα αυτά. Σας, σας ευχαριστούμε λοιπόν που φροντίζετε τις σχέσεις σας μαζί μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τις απαντήσεις σας και για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ. Uh, Συνάδελφοι, θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Παρακαλώ, έχετε έτοιμε τι κάρτε σα. Αν δεν έχετε τις κάρτε σα, πείτε το μου σα παρακαλώ. Συνάδελφοι, αν κάποιος δεν έχει την κάρτα του μαζί σας, παρακαλώ πείτε το μας και θα καταγράφουμε την ψήφο σας διανατάσεως. Ε, συνεχίζουμε λοιπόν με το θέμα 8. Πρώτη ψηφοφορία για επί το κείμενο που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο των διοργανικών διαπραγματεύσεων. Πρόκειται για το κείμενο στο οποίο καταλήξαμε στη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων ε, στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Είναι ένα από τα βασικά θέματα που ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας και χαίρομαι που επετεύχθη σχετικά γρήγορα αυτή η άτυπη συμφωνία. Ε, προτού προχωρήσουμε στην πληροφορία, η συγγήτρια κυρία Χολμάιρ θέλει να τοποθετηθεί. Παρακαλώ. Πάρα πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε την ε, Κατερίνα, αλλά και με όλες τις πολιτικές ομάδες. Πραγματικά η συνεργασία μας ήταν εξαιρετική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Γκάι, ο οποίος μας ε, συνόδευσε πραγματικά με εξαιρετικό τρόπο από πλευράς γραμματείας της ΛΥΜΠΕ. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Προεδρία του Συμβουλίου για την ε, εξαιρετική συνεργασία τους, την επικοδομητική τους στάση και την προσπάθεια να εξευρεθούν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις. Ήταν ε, μεταξύ άλλων και ο λόγος για τον οποίο καταφέραμε να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο ισορροπημένο κείμενο το οποίο μάλιστα καταφέραμε να το επιτύχουμε και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Συζητούμε λοιπόν ε, και ψηφίζουμε μάλλον επί του κειμένου στο οποίο κατέληξαν οι διοργανικές ε, ψηφοφορίες. Ε, ονομαστική ψηφοφορία ψηφίστε παρακαλώ. Ένας ψηφοφορίας. Sorry, um, E Το ΕΛΚ έχει δύο ε, υπεράριθμους ψηφίσαντες. Εντάξει, τώρα είναι εντάξει. Τέλος της ψηφοφορίας. 37 υπέρ, 4 ψήφοι κατά, 7 αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Και πάμε κατευθείαν στην επόμενη ψηφοφορία που είναι το σχέδιο γνωμοδότησης για την ετήσια έκθεση του 2015 για την προστασία της, των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολέμηση απάτης. Κυρία Τζίνη είναι εισηγήτρια. Αν θέλει το λόγο τον έχει, αλλιώς περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Πάμε στην ψηφοφορία. Θέλω απλώ να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, συνεισηγητές και όσους συνεργάστηκαν μαζί μου για αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Ευχαριστούμε κύριε Κίνιτσι. Πάμε στην ε, τροπολογία 1, παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Sorry, you voted. Could somebody record? Um... μπορεί κάποιος να καταγράφει την ε, ψήφο της κυρίας Μπενόβα. Μπορείς, σε παρακαλώ, να καθίσεις ε, δίπλα για να χρησιμοποιήσεις το... Όχι, δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Εντάξει, θα καταγράφουμε την ψήφο σου. Εδώ χειροκίνητα. Δεν λειτουργεί το μηχάνημά σας, κύριε Κουρίκα. Όχι, εντάξει, λειτουργεί. Εντάξει. Τροπολογία 2. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 3. Ένας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 4. Ένας ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 5. Ένας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 6. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Έναρξη ψηφοφορίας. Ε, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Η ε, έναρξη ψηφοφορίας. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 13. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 14. Έναρξη ψηφοφορία. Πέραση της προφορίας... Απορρίπτεται. Συμβαστική 2, πρώτο τμήμα, έναρξη ψηφοφορίας. Πέραση προφορίας... Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, έναρξη προφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3, έναρξη ψηφοφορίας. πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 23, Ένα ψηφοφορίας. Πέρας εγκρίνεται. Ψηφοφορία από το κειμένο όπως τροποποιήθηκε. Έναρξη ψηφοφορίας. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 42 υπέρ, 3 κατά τρεις αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, την κυρία Τσίνιτσι. That is the end of time, colleagues, and we... Φτάσαμε στο τέλος των ψηφοφοριών, συνάδελφοι. Διάφορα δεν έχουμε. 8 Δεκεμβρίου επόμενη συνεδρίαση. Κυρίσω τη λήξη της σημερινής μας συνεδρίασης.